Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, με συγχωρείτε, πρέπει να κάνω τηλεφώνημα και άρχισα Χαιρετίζω τον παλιό και τον νέο μας επιτροπό. Σας γνωρίζουμε, αλλά χαιρόμαστε που έχεις αναλάβει θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας και σε ευχαριστώ για την παρουσία σου και χαιρετίζω εξίσου θερμά και τους συναδέλφους από το Ελεκτικό συνέδριο, τον κύριο Λαζάρο. Σας είδαμε και χθε την κυρία Τότελμουντ, Γκρέγουαρ και Εύα Λίνστρομ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει τόσο πολύ άριθμοι και χαίρομαι που θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε για, την, για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και για τα διδάγματα που έχετε εξαγάγει από την εξέτασή του. Καταρχάς, να δώσω το λόγο στα τέσσερα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Αν κατάλαβα καλά, θα ξεκινήσει ο κύριος ε, Λαζάρου, έτσι δεν είναι. Μάλιστα, παρακαλώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Επίτροπε Χάν, καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Χάν που είναι επίτροπο για τον προπολογισμό σε αυτή τη νέα του θητεία. Προπολογισμό και διοίκηση. Οι συνάδελφοι μου και εγώ προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του για να συμβάλλουμε στι προσπάθειε του, τόσο ώστε να δαπανάται σωστά ο προπολογισμό με βάση του κανόνε και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στου πολίτε Και θέλουμε η Επιτροπή να παρουσιάζει σωστά τι ε, δραστηριότητε τη για να μπορούμε και εμεί να κάνουμε τον ελέγχο. Ο Επίτροπος Χάν εκπροσωπεί συνολικά την Επιτροπή γιατί συζητάμε τα οριζόντια κεφάλαια. Συμμετέχω σε αυτήν την ακρόαση μαζί με την κυρία Τάτλμπομ που είναι υπεύθυνη για το κεφάλαιο 2 για την οικονομική και νομισματική διαχείριση ο κύριος Γκρέγουαρ που είναι για το κεφάλαιο 3 πώς θα έχουμε αποτελέσματα από τον προϋπολογισμό και η κυρία Λίνστρομ που είναι για το 4 για τα έσοδα ως μέλος για την ετήσια έκθεση για το κεφάλαιο 1 λοιπόν που δίνει και την ε, δήλωση αξιοπιστία του ελεκτικού συνεδρίου είχα την ευκαιρία να συζητήσω τι παρατηρήσει μα ενώπιον τη Επιτροπή σα στις 8 Δεκάτου. Η δήλωση αξιοπιστία είναι καθαρή για του λογαριασμού και τα έσοδα του 2018 και για τρίτη χρονιά κατά σειρά. Έχουμε επιφυλάξει για τι δαπάνε ιδιαίτερα δαπάνε υψηλού κινδύνου, επιστροφέ, και αυτό συμβάλλει στην, στο ουσιώδες ποσοστό σφαλμάτων. Θέλω να είμαι σύντομος για να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση και για τους άλλους συναδέλφους από το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τότελμπου. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το κεφάλαιο 2 τη ετήσια έκθεση 2018 του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ο κύριο στόχο μα είναι, είναι να εξετάσουμε και κατά πόσο η διαχείριση λειτουργεί σωστά και αν γίνονται σωστά εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τονίσουμε τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια. Ασχολούμαστε κυρίως ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Δηλαδή, Ακόμη και αν δεν έχει οικονομικό αποτέλεσμα ένα σφάλμα, μπορεί να έχει ουσία γιατί είναι σημαντική για τα πορίσματά μας. Ακόμη και αν αφορά ένα μικρό ποσό. Από τη φύση του έχει ουσία. Τα θετικά. Στον προπολογισμό του 18 η Ένωση και οι υποχρεώσεις και οι πληρωμές αξιοποιήθηκαν σχεδόν πλήρως. Αλλά σε τέσσερις τομείς υπάρχουν κίνδυνοι για τον προπολογισμό που εντοπίσαμε. Πρώτος, αφορά ε, τις αξιώσεις AC. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Στο τέλος 2018, μόνο 27% του συνόλου δαπανήθηκαν προς τα κράτη-μέλη, ενώ το 2011 ε, ήταν, ήταν 33%. Άρα το ποσοστό απορρόφηση από τα κράτη-μέλη το 2018 μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Κροατία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Η Φινλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης. Η αύξηση προβλημάτων με τις υποχρεώσεις είναι κάτι που τονίζουμε στο κεφάλαιο 2. Η καθυστέρηση στην εφαρμογή των χρηματοδοτήσεων αυξάνει τα RAL, τα Resta Liquide, που είναι 81 δις για το 2018. Όπως βλέπετε εδώ, το RAL έχει αυξηθεί συνεχώς από το 2017 και προβλέπεται το 2023 να φτάσει στα 340 δις. Θα έχουμε πρόβλημα ρευστότητας και μπορεί να μην έχουμε επαρκής ε, πιστός υποχρεώσεων για το επόμενο πολιτές πλαίσιο. Αν εξετάσουμε λίγο βαθύτερα το θέμα αυτό, θα συστήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση για τις υποχρεώσεις στα πρώτα χρόνια του επομένου πολιετούς πλαισίου και να κρίνονται τα πολιτή προγράμματα εγκαίρως. Η αύξηση των εγγυήσεων μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τον προπολογισμό. Οι εγγυήσει είναι για να χρησιμοποιήσουμε και εξωτερικούς πόρους για να έχει περισσότερη επίπτωση ο προπολογισμό. Η αύξηση των εγγύσεων τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίω στην αύξηση του ΕΦΣΥ και του EFSD, δηλαδή στην αύξηση των εγγύσεων που δίνονται στα πλαίσια αυτών των ταμείων. Όπω βλέπετε εδώ στο PowerPoint, η έκθεση θα αυξηθεί σταδιακά όσο γίνονται πληρωμές. Στο τέλος του 2018 οι εγγύησεις ήταν 92,8 δις. Οι εγγύησεις καλύπτουν τις απώλειες που προβλέπει η Επιτροπή και στο επόμενο πολιτές πλαίσιο αυτές οι εγγυήσεις θα ε, είναι σε ένα κοινό ταμείο προβλέψεων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε την ε, έκθεση σε εγγύησεις και επίσης να έχουμε μία σόφρονα μεθοδολογία με βάση τις αναγνωρισμένες καλές πρακτικές. Τέταρτο και τελευταίο που εκθέτει τον προπολογισμό σε κίνδυνο είναι ότι η Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαφορετικούς λογιστικούς κανόνες παρά το, ότι είναι τμήμα του θεσμικού μας πλαισίου δεν είναι θεσμός της Ένωσης έχει διαφορετικούς κανόνες ε, διαχείρισης και διακυβέρνησης και όπως βλέπετε στο 4 οι πληρωμές από τον προπολογισμό της Ένωσης στον προπολογισμό της Τράπεζα Επενδύσεων έχουν τα τελευταία χρόνια. Συνολικά 40,7 δις δεσμεύθηκαν από τον προβλημό της Ένωσης για την ε, Τράπεζα Επενδύσεων και αυτή η τάση θα αυξηθεί και στο επόμενο πολίτες πλαίσιο. Ο ρόλος της ε, Τράπεζα Επενδύσεων αυξάνεται. Οι νέες επενδύσεις του EFSD θέλουν να ε, μοχλεύσουν 650 δις και ο προπολογισμός της Ένωσης θα δώσει εγγύησεις 38 ε, δις. Η κατάσταση αυτή μας οδηγεί στο να πούμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να δώσει στις αρχές ελέγχου του προπολογισμού συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς κατανέμονται οι πόροι από τον προπολογισμό της Ένωσης που πηγαίνουν στα χρηματοδοτικά μέσα που ελέγχονται από την, ε, που μάλλον που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Μεδίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη Γκρέγκορ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, θα προσπαθήσω εν συντομία να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο 3 που επικεντρώνεται στις ε, επιδόσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τέτοιο κεφάλαιο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις αιτήσεις εκθέσεις μας το 2010 και έκτοτε προσπαθούμε να αξιολογούμε τις επιδόσεις επιλεγμένων προγραμμάτων το 2014, ε, το 2014 ξεκινήσαμε την αξιολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων με ε, συγκεκριμένα κεφάλαια που αφιερώνονταν. Το, στη συνέχεια όμως ε, το 2016 προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε με πια οριζόντια προς οπτική αξιολόγησης ε, κοιτάξαμε τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για την λήψη αποφάσεων και για το 2018 αναλύσαμε ποιες ήταν οι επιδόσεις και οι, και οι αντίστοιχοι δείκτες και τι μας ε, λένε. Εξολογήσαμε 22 συνολικά προγράμματα και δείκτες που αναφέρονται στα, στις δηλώσεις των προγραμμάτων, στα σχέδια προπολογισμού του 2019 και όλα αυτά δημοσιεύτηκαν ε, για πρώτη φορά τον Μάιο του 2018. Μια επισκόπηση δηλαδή ε, των επιδόσεων των προγραμμάτων. Ήταν ένα έγγραφο πολύ χρήσιμο για να μας ε, δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να αναλύσουμε καλύτερα τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επίσης, Αναλύσαμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, όπως βλέπετε εδώ στο τμήμα 1α του κεφαλαίου 3, στο τμήμα β ε, καταλήξαμε σε μια γνώμη ότι τα αποτελέσματα δεν σκιαγραφούν πάντοτε την πραγματική πρόοδο. Γιατί, για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, πολλοί δείκτες δεν είχαν επιλεγεί σωστά, γιατί 60% των δικτών από την δική μας ε, οπτική είναι ε, δείκτες input-output και κάποιοι δεν συνδέονται σαφώς με τις δαπάνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν καλύπτονται ορισμένες πτυχές από κάποιους δείκτες. Επίσης, είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς την ε, πρόοδο για κάποιους δείκτες, για συγκεκριμένους δείκτες. Για το 44% των δικτών δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάλι για διάφορους λόγους, γιατί δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι στόχοι, δεν υπήρχαν ε, τιμές βάσης ή επειδή ακολουθούνταν διαφορετική μεθοδολογία με διάφορους δείκτες στο πέρασμα του χρόνου. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ και στα άλλα δύο τμήματα του κεφαλαίου 3, που είναι μια επισκόπηση των συστάσεών μας για το 2018. Είχαμε 184 συστάσεις ε, στους ε, ελεγχόμενους, η πλειονότητα των οποίων έγινε πλήρως αποδεκτή, 62% το 10... των ε, συστάσεων, το 94% μάλλον ε, των συστάσεων μας ε, έγινε δεκτή, μόλις το 6% δεν έγινε δεκτό, 6%. Επίσης παρακολουθήσαμε και την εφαρμογή των συστάσεων μας. Φέτος επικεντρωθήκαμε στην εφαρμογή των συστάσεων του 2015 και εδώ η πλειονότητα των συστάσεών μας διαπιστώσαμε ότι είχε εφαρμοστεί πλήρως. Αυτά από εμένα και σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την ευσύνοπτη παρουσίαση των ε, στοιχείων σας για να μας μείνει και χρόνος για να μπορέσουμε να σας, βάλουμε, να σας υποβάλουμε και ερωτήσεις. Η κυρία Λίντστρομ έχει το λόγο τελευταία εκ των τεσσάρων προσκεκλημένων μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κύριε Χάν, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο 4 εν συντομία. Εδώ και πολλά χρόνια τα έσοδα του προπολογισμού δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό τμήμα. Πλέον όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χρηματοδότηση της Ένωσης, πλέον τα έσοδα ε, ε, έχουν μεγάλη σημασία και αυτή αναγνωρίζεται και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις αιτήσεις εκθέσεις μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, οπότε θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία στην παρέμβασή μου. Πρώτον, τι διαπιστώσαμε. Είδαμε ένα δείγμα 55 εντολών ανάκτησης, αξιολογήσαμε τα συστήματα ελέγχου τη Κομισιόν και των κρατών μελών. Φέτος επισκεφτήκαμε την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία και τέλο κάναμε μια εκτίμηση για τι ε, ετήσιε εκθέσει ε, τη Eurostat και τη γενική διεύθυνση προπολογισμού. Βλέπουμε ότι, βρήκαμε ότι το σφάλμα ε, στις, στα έσοδα δεν ήταν υλικό, ωστόσο στους παραδοσιακούς ε, ιδίους πόρους και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη ήταν τα συστήματα ελέγχου μόλις εν μέρη αποτελεσματικά. Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία διαπιστώσαμε αδυναμίες ε, όσον αφορά την, ε, τη διαχείριση των ε, λογαριασμών Β και την ίσπραξη των δασμών. Στην Ισπανία επίσης διαπιστώσαμε προβλήματα στο σύστημα τήρησης λογαριασμών. Επίσης διαπιστώσαμε προβλήματα στις δηλώσεις της Κομισιόν, των κρατών μελών προς την Κομισιόν σχετικά με την υποβολή των παραδοσιακών ιδίων πόρων. Ε, εδώ προτείνουμε να γίνεται καλύτερη ανάλυση κινδύνου και σε, σε επίπεδο κράτους μέλους. Επίσης, ε, καλούμε ε, τις εμπλεκόμενες αρχές να ελέγχουν σε μεγαλύτερο βάθος ε, ασυνήθιστες αλλαγές που διαπιστώνονται στις αιτήσει δηλώσεις. Εμείς πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε μόνο αυτά που ήδη έχουν ενταχθεί στους λογαριασμούς και αν αυτά είναι σωστά. Αν θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί περισσότεροι δασμοί, περισσότερο ΦΠΑ, αν υπάρχει απάτη για παράδειγμα, αυτά τα εξετάζουμε σε ειδικές εκθέσεις που συντάσσουμε. Έχουμε ε, επίσης και κάποιες συστάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα όσον αφορά την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Και για το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, έχουμε υποβάλει μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη ε, και διαπιστώνουμε ότι και οι αρχές των κρατών μελών και οι ενωσιακές αρχές ε, είναι αδύναμες ε, όσον αφορά τον έλεγχο των προβλημάτων ή των κινδύνων που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τρίτον, να σας πω κάποια λόγια για τις νομοθετικές προτάσεις και εξελίξεις που υπήρξαν ε, σε σχέση με τα έσοδα και για το μέλλον. Το 2018 η Κομισιόν πρότεινε ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων και εμείς γνωμοδοτήσαμε επί του συστήματος αυτού, της πρότασης δηλαδή της Κομισιόν. Εγώ ήμουν υπεύθυνη η διαδικασία βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση βεβαίω και ε, σκοπό τη Κομισιόν είναι η απλοποίηση του συστήματο και η ένταξη νέων ε, ιδίων πόρων που θα συνδέονται με νέου τομεί πολιτική. Εμεί είχαμε ήδη εκφράσει τι ανησυχίε μα ε, για το νέο αυτό σύστημα ιδίων πόρων για την εταιρική βάση και την φορολόγηση αυτής, για, το, για, τις πλαστικές και το ε, σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ε, δεν, εμείς είχαμε διαπιστώσει ε, και είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι προτάσεις εξακολουθούν να είναι αδύναμες και δεν συμβάλλουν στην απλοποίηση του συστήματος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα αν τα ζητήματα που εξετάζουν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Όλαφ και σε ειδική μας έκθεση καλέσαμε, σημειώσαμε την ανάγκη να αποκτήσει ο Όλαφ ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά την ίσπραξη και την ανάκτηση ε, ποσών, ε, ιδίως στους τομείς όπου υπάρχει διασυνοριακή ε, απάτη. Επίσης η Ευρωπαϊκή Συγγελία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και στις εκθέσεις Κομισιόν περιλαμβάνονται μια σειρά από στόχοι, οι οποίοι επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να κατατείνουν πάντοτε στην βελτίωση του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ κυρία Λίνστρομ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια είχα τη χαρά να κάνω τακτική ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας και χαίρομαι που θα συνεχίσω και στην επόμενη πενταετία. Κάποιες φορές ε, μπορεί να είχαμε και διάσταση απόψεων για κάποια θέματα, αλλά έχουμε ένα κοινό στόχο να εξασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδει προστιθέμενη αξία, αντιμετωπίζει τις ε, προκλήσεις και ε, δαπανούμε καταλήλως τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και φυσικά μεταξύ των κρατών μελών και φυσικά και με το ελεγκτικό συνέδριο. Γνωρίζω επίσης ότι εσείς κυρία Πρόεδρε και αρκετοί από τους συναδέλφου ε, είστε στην αξιοσημείωτη ε, θέση να εξασφαλίσετε ότι τα σφάλματα του παρελθόντος ε, θα μετατραπούν σε αποφάσεις βάσει κατάλληλης ενημέρωσης και θα δαπανούνται κατάλληλα ε, τα κονδύλια του προπολογισμού. Και αυτά όλα σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν το έργο μα. Όπω εξήγησε ο κύριο Λαζάρου και οι συνάδελφοί του, και ευχαριστώ και πάρα πολύ για τη δουλειά του και την ε, καλή μα συνεργασία, πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο εκκίνησης με σαφή άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου και ε, πολύ χαμηλότερα ποσοστά ασφάλματος για τις δαπάνε από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε επίσης ε, πολύ υψηλότερη στόχευση για τις επιδόσεις των ε, προγραμμάτων δαπανών και αυτή είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Σήμερα με τη νέα μου ιδιότητα ε, ω επίτροπο για τον προπολογισμό και τη Διοίκηση θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιε από τι προκλήσει και τι ευκαιρίε που μα προσφέρονται. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός βελτιώνει τη ζωή των ε, Ευρωπαίων πολιτών και να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά τους, να δημιουργήσουν νέα προγράμματα να ανοίξουν νέε αγορέ, Υποστηρίζουμε πρόσβαση σε ε, υψηλής σε βριζονικά δίκτυα και σε σπίτια και σε επιχειρήσει, ενίσχυση των νέων τεχνολογιών και συμβάλλουμε ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν εκεί που επιθυμούν και να μην υποχρεώνονται, για παράδειγμα, να μετικήσουν ε, σε άλλες ε, περιοχές. Επίσης, ε, ε, προχωρούμε προγράμματα καινοτομίας ε, στην υγεία για να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες. Για παράδειγμα, η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θα αποσχολήσουν την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάποια παραδείγματα και μόνον. Αλλά όταν μιλώ με τους πολίτες, πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τι αποκομίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζουν πώς οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό αλλάζουν την καθημερινότητά Επομένως, η κοινή πρόκληση και υποχρέωσή μας είναι να τους εξηγήσουμε λίγο καλύτερα ε, τα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και να τους βοηθήσουμε να εκτιμήσουν την προστιθέμενη αξία και τη σημασία των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, πρέπει να αποδείξουμε ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε νέε και καλύτερε επιλογέ όταν ένα πρόγραμμα δεν αποδίδει όπω θα περιμέναμε. Ο ΩΣΑ επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα προηγμένο πλαίσιο για την μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων για τι επιδόσει με σαφεί στόχου και δείκτες, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε. Και επ' αυτού πρέπει να αναρωτηθούμε εάν έχουμε θέσει σαφεί ε, στόχου και αντικειμενικού σκοπού ε, με αντικειμενικού δείκτε, αν συλλέγουμε τα πλέον κατάλληλα στοιχεία και πληροφορίες και εάν τα παρουσιάζουμε με τον πλέον χρήσιμο τρόπο και τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις πολιτικές μας καλύτερες. Θέλουμε να σας προσφέρουμε ε, εσάς και στους συναδέλφους σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σαφή βάση για τις επιλογές του μελλοντικού προπολογισμού και τη δυνατότητα επαλλαγής για, τον προηγούμενο, για τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Προβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας και με το ελεγκτικό συνέδριο για τον τομέα αυτό. Υπάρχει ένα περίπλοκο περιβάλλον με πληθώρα εταίρων και ε, συνδεδεμένων ε, χωρών και φυσικά διεθνών οργανισμών. Οι δικαιούχοι βρίσκονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια συχνά δαπανώνται πολύ μακριά από τις Βρυξέλλες. Σε ένα τέτοιο λοιπόν σύνθετο περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που διαχειρίζονται τα κονδύλια επιτόπου θα κάνουν όσα πρέπει βάσει των κανόνων μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και του υπόλοιπου εταίρου, συνεχίζουν να εργάζονται προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνο και όπου δει ε, να λαμβάνουν μέτρα για τα προβλήματα που διαπιστώνονται. Για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε υψηλά πρότυπα για την διαχείριση και να επικεντρωνόμαστε στους βασικούς κινδύνους. Βρέσκω ότι τα ποσοστά σφάλματος είναι ένα σύστημα δικτών που μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά είναι απλώς δείκτες και απλώς μας δίνουν τμήμα της γενικότερης εικόνες. Το ελεγκτικό συνέδριο θέλει να ε, εξυγχρονίσει τη δήλωση ε, ε, και την προσέγγιση για τα διορθωτικά ταμεία. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το ηλεκτρικό συνέδριο στην προσπάθειά του. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε πώ μπορούμε να συνεχίσουμε από τα διδάγματα που αντλήσαμε και να λάβουμε τα ε, μέτρα που απαιτούνται και να επεκτήσουμε την ε, προσέγγιση μα και σε άλλα σκέλη του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Εγώ δεσμεύομαι για αυτή τη διαδικασία και είμαι βέβαιος ότι η κοινή μας προσπάθεια θα αποφέρει καρπούς. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε αξιόπιστες πληροφορίες, αν είναι και επαρκούς ποιότητα. Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι να βελτιστοποιήσουμε την ε, ε, απορρόφηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και να ε, επικεντρωθούμε στους ε, πιο βασικούς τομείς. Δεν θα διστάσουμε να συζητήσουμε και λεπτά ζητήματα όπως τη σύγκρουση συμφορώντων ή το κράτος δικαίου. Να τονίσω ότι τα σφάλματα δεν σημαίνουν ότι σπαταλούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή χάνονται, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ε, μηδενική ανοχή στην απάτη και εγώ θέλω να ε, εργαστούμε περισσότερο προκειμένου να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η συνεχής αναθεώρηση του κανονισμού ε, της Όλαφ, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι όλα βήματα προς σωστή κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει αυτό το δρόμο. Επίσης θα επικεντρωθώ στην προστασία των ε, χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών και ε, έχουμε και τους δύο φορείς που έχουν την εντολή να καταπολεμήσουν την απάτη, την Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν καλύτερη προστασία του ευρωπαϊκού ε, προπολογισμού, δίωξη των εγκληματιών, των και ανάκτηση των κονδυλίων. Να πω και δύο λόγια για την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αποδίδει καταλήλωση η διοίκησή μας, επομένως εγώ δεσμεύομαι για μια επιτροπή η οποία θα κάνει μια αλλαγή στα ψηφιακά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λύσεις ε, ψηφιακής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των βασικών πολιτικών και της απλής διοίκησης. Αυτό θα οδηγήσει και σε αποδοτικότητα προ το κόστο, αλλά θα δημιουργήσει και σε συντονισμό. Έχουμε κάνει κάποια βήματα προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά η πρόκληση είναι να εξυγχρονίσουμε και να εκλογικεύσουμε το ψηφιακό μας ε, ε, σύστημα με συγκεκριμένο και ε, λογικό τρόπο. Και εδώ θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτελέσει το καλό παράδειγμα, να ε, υποστηρίξει τα κράτη-μέλη για την μετατροπή του δημόσιου τομέα, ώστε να είναι έτοιμοι για την ψηφιακή εποχή. Πρέπει να συνεργαστούμε και νομίζω ότι ο βασικός όρος θα είναι διαλειτουργικότητα. Είναι μία από τις βασικές προκλήσεις και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τουλάχιστον να βοηθήσουμε ώστε σταδιακά τουλάχιστον να να εφαρμοστεί αυτό. Να έρθω και στο τελευταίο σημείο, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις, ε, έχουμε και τη διαδικασία της απαλλαγής. Ε, όλα αυτά ε, έχουν μεγάλη σημασία για τις δομές και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και της χρηματοδότησης. Πρέπει να κάνουμε επιλογές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο για το μέλλον, πρέπει να υπάρχουν πόροι γι' αυτό. Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στις επιδόσεις, θα πρέπει να υποστηρίξουμε προγράμματα και κατάλληλου δείκτε επ' αυτού. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμόρφωση με τους κανόνες και να μειώσουμε τα ποσοστά φάλματα, τότε θα πρέπει να είμαστε υπέρ απλών κανόνων. Ήδη λάβαμε υπόψη ε, πολύ καλέ συμβουλέ που λάβαμε από το ελεγκτικό συνέδριο, όταν ε, καταρτήσαμε τις προτάσεις. Τώρα πλέον χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά προγραμμάτων θα είναι ακόμα καλύτερη από αυτά που έχουμε τώρα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και η Φιλανδική Προεδρία είναι στη μοναδική θέση να μπορέσει να θέσει το βηματισμό για τη συμφωνία. Είναι πολύ λεπτή η διαδικασία, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου ε, είναι ίσω ε, το αποφασιστικό βήμα για το πώ θα προχωρήσουμε οι διαπραγματεύσει για να έχουμε έναν ισορροπημένο σύγχρονο προπολογισμό για την επόμενη επταετία. Τώρα πλέον να αποφασίσουμε και το συντομότερο θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει γιατί έτσι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αυτό θα βοηθήσει να ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο για να έχουμε συνένεση. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω και πάλι λογική, ισορροπημένε θέσει και ένα βασικό κοινό στόχο ε, για τα τρία θεσμικά όργανα. Να εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κατάλληλα μέσα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, αγρότε, φοιτητέ, εργαζομένους, μικρομεσαίε επιχειρήσεις, επιχειρηματίε. Θέλουμε να διδαχθούμε από το παρελθόν για να βελτιώσουμε το μέλλον. Επομένω, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα για να εξασφαλίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα αντιμετωπίζει τι βασικέ μα προτεραιότητε για το μέλλον και ότι θα σεβαστούμε τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνεια και λογοδοσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε μαζί αυτό το ταξίδι, μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και πολλέ νέε ιδέε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλε αυτέ οι ευκαιρίε κατά τη διάρκεια τη θητεία μα και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε πιο απλού και πιο εύρωστου κανόνε που ταυτόχρονα θα βοηθήσουν να εξοπλίσουμε και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για τους πολίτες μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας κάνουμε και ερωτήσεις γιατί θα είμαι εγώ η συγγήτρια. Να ξεκινήσω με τα ε, γάλ, το υπόλοιπο προς εκαθάριση, που αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα. Θέλουμε να μην υπάρχουν κίνδυνοι για την εκτέλεση του προπολογισμού και αυτά τα γάλα είναι χρέη γιατί υποβάλλονται οι αποδείξεις στα κράτη-μέλη για το επόμενο πολιτές πλαίσιο όπως μας είπε το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει κίνδυνος κρίσης πληρωμών τι μέτρα προβλέπει η Κομισιόν για να αποφευχθεί αυτή η κρίση το 2021 και 2022 που θα είναι τα δυσχερέστερα έτη. Δεύτερον, από την πείρα του παρόντος πολιετούς ε, πλαισίου υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για το επόμενο. Για παράδειγμα ο κανόνας 1 συν 3. Μήπως πρέπει να αλλάχθεί για να μην προκύπτουν οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα. γιατί το 0,99% είναι υποχρεώσεις τα προγράμματα ξεκινάνε με μεγάλη καθυστέρηση και αναμένουμε ότι και στο επόμενο θα είναι μεγάλη καθυστέρηση και επειδή υπάρχουν αυτοί οι κανόνες 1 συν 3 τα παλιά προγράμματα λήγουν πολύ αργότερα οπότε μπερδεύονται οι δομές των πολιετών ε, προοπτικών. Τα νέα προγράμματα καλύπτουν το παλιές δαπάνες και αντίστροφα. Θα έχουμε όλο και δυσχερέστερη κατάσταση όσο προχωράει η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεύτερον, που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είπαμε που είναι μεγαλύτερη κίνδυνο από πλευρα... κίνδυνη από πλευράς ε, τάξης μεγέθους. Και το πρόβλημα λοιπόν για τους ίδιους πόρους είναι η απάτη του ΦΠΑ. Ποικίλουν τα νούμερα, αλλά επειδή συζητάμε για τον προϋπολογισμό 220, εμείς θεωρούμε ότι θα είναι 500 εκατομμύρια. Και μετά έρχεται η Europol και μας λέει ότι θα είναι πολλά, πολύ περισσότερα. Οπότε παραδέχομαι ότι αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι για τρεις μέρες για αυτά τα 500 εκατομμύρια και ε, μετά η Ευρωπόλ μας λέει ότι είναι 5 δις. Θα μπορούσε να μας πει και 80 και 90. Είναι πολύ διαφορετική η τάξη μεγέθους. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά στο μέλλον, στο μέλλον ούτω ώστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν διαμεθοριακά αυτά τα θέματα. Πού είναι οι αδυναμίες ε, στην ίσπραξη του ΦΠΑ. Πολλά προβλήματα ηλεκτρονικού εμπορίου προκύπτουν. Θα πρέπει ίσως να το συζητήσουμε το θέμα του ΦΠΑ εκτενέστερα γιατί είναι τεράστιο θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα. Για τα τελωνιακά υπήρξε ειδική έκθεση του συνεδρίου όπου τονίζονται οι αδυναμίες του συστήματος τελωνίων μας και ότι αυξάνεται η απάτη για κάποιες κατηγορίες αγαθών και μπορεί να έχουμε σημαντικές ε, σημαντικά ποσά απολειών, εάν δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για παράδειγμα. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε πώς θα καλύψει αυτά τα κενά, αυτές τις δυσχέρειες που τα, τις έχουμε χρόνια και χρόνια, πώς θα ενισχύσουμε τα τελωνία και κυρίως τη συνεργασία μεταξύ των διαφορών υπηρεσιών τελωνίων. Τέταρτον, Βεβαίω και οι συνάδελφοι μετά θα κάνουν ερωτήσει γιατί για τον ΦΠΑ είναι πολύ ασαφή η Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη μπορεί να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Αυτό το γνωρίζω. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε πού είναι τα εντονότερα προβλήματα. Να μου πείτε πού εντοπίζετε τους μεγαλύτερους κινδύνους. Τώρα κάτι εντό αγωγικών μικρότερες σημασίες. Στο πολίτικο διάβασα ότι η Κομισιόν ε, προβλέπει περισσότερους πόρους, κατά 50% περισσότερους πόρους για πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα για τους ε, ηθήνοντες. Τι είναι αυτό, είναι φυσιολογική αύξηση. Είναι λάθος αυτό που μας λέει το πολίτικο. Εάν δεν είναι δυνατόν να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις τώρα, παρακαλώ να ε, μου αποστείλετε γραπτές απαντήσεις. Και τελευταίο. Συνοχή και γεωργία. Έχουμε τη νέα έκθεση για την τσεχική δημοκρατία. Και ακούμε και διαβάσαμε και στην εφημερίδα New York Times. Μήπως υπάρχει θέμα αρπαγής γης και άλλων καταχρήσεων στη χρήση πόρων. Πόρων συνοχής. γιατί υπάρχουν κάποιες ε, ολιγαρχικές δομές από ό,τι φαίνεται. Στόχος μας δεν είναι να ενισχύουμε αυτές τις ολιγαρχικές δομές, τους γεωκτήμονες, αλλά να ωφελούνται περισσότεροι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά διαβάζουμε εδώ τίτλους και μάλιστα χθες σε άρθρα. Και μετά διαβάσαμε την έκθεση αυτή στο ίντερνετ την ειδική έκθεση για τα θέματα αυτά. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί ε, επισήμως δεν την έχουμε λάβει ακόμη, αλλά υπάρχει στο ίντερνετ. Εγώ είμαι τη Επιτροπής ε, Προπολογισμών. Ε, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να μην την έχουμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τη συζητάμε, αλλά αφού είναι στο ίντερνετ μπορούμε να τη διαβάσουμε. Τι είναι αυτά. Εντυπωσιακά για να το πω με ήπιο τρόπο. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε πλήρως σήμερα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πώς θα ενισχύσετε τα μέτρα για να σταματήσουν αυτά τα πράγματα, που δεν είναι πια μεμονωμένα. Επαναλαμβάνονται και δημιουργούν δυσπιστία στον πληθυσμό για την εργασία μας. Δημιουργούν την εντύπωση ότι οι πλούσιοι παίρνουν τα πολλά και οι υπόλοιποι ψίχουλα. Τι είναι αυτά. Εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σας παρακαλώ να τοποθετηθείτε και για αυτά. Καταλαβαίνω, αν δεν μπορείτε να μπείτε στις λεπτομέρειες τώρα, να τα πούμε αργότερα. Ich habe mir erstmal. Okay, exklusive Beantwortung, gerne. Ωραία, να απαντήσω αποκλειστικά σε εσά. Κοιτάξτε μα αυτό είναι προνόμιο των εισηγητών. Πρώτη ερώτηση. Τα υπόλοιπα προς εκαθάριση. Ασχολήθηκα για πρώτη φορά με το θέμα αυτό και με εκνευρίζουν αυτά τα στοιχεία. Συζήτησα με τους συνεργάτες μου, αλλά αυτοί είναι πιο ήρεμοι. Μου είπαν ότι άμα δούμε τη χρονική εξέλιξη είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία ε, αυξάνονται κάπως αλλά ο φόβος να υπάρξουν πραγματικά προβλήματα ρευστότητας δεν είναι πολύ υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος. Με ρωτήσατε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στο μέλλον. Τι διδάγματα εξάγουμε από το παρόν πολιτές πλαίσιο για το μέλλον, για το επόμενο. Αναφερθήκατε στο κανένα εν συν 3. Νομίζω ότι ο Επίτροπος για τα περιφερειακά θέματα δεν ήταν πολύ ικανοποιημένος από αυτόν τον κανόνα, αλλά έπρεπε να τον τηρήσουμε για μετά από πίεση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα προτιμούσαμε το νισιν 2. Αλλά μας υπόθηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθούν κάποια προγράμματα. Δηλαδή, οι χώρες που έχουν δυσχέρειες εφαρμογής πίεσαν για να έχουν ένα χρόνο παραπάνω. Και αυτό προκαλεί αυτές τις καθυστερήσεις. Αυτή την ε, συσσόρευση χρεών. Το άλλο έχει να κάνει και ότι είναι αποφασιστικό πότε αποφασίζεται το πολιετές πλαίσιο για να μπορέσει να αρχίσει η εφαρμογή της νέας περίοδου. Αν θυμάστε, την τελευταία φορά η απόφαση για το παρόν πολυονομικό πλαίσιο ελήφθη στις 13 Δεκεμβρίου του 2013 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου του 2014. Ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και από τη μια στιγμή στην άλλη. Έπρεπε να αποφασιστούν οι κανονισμοί, να εγκριθούν τα προγράμματα. Δηλαδή, κουβαλάμε την καθυστέρηση. Τώρα, από τη θετική πλευρά, είχαμε εισαγάγει τότε την υποχρέωση να μας υποβάλουν στρατηγικές για τους διάφορους τομείς στα κράτη-μέλη ως προϋπόθεση απελευθέρωσης των πόρων. Θυμάμαι ότι ο Περιφερειακός Επίτροπος αντιμετώπισε πολλές επικρίσεις σε κάποια κράτη-μέλη ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουμε περιφερειακά αεροδρόμια κτλ αλλά έκτοτε δεν έχω ακούσει τόσο πολλές επικρίσεις γιατί απαιτήσαμε από τα κράτη-μέλη να μας υποβάλουν πρώτα μία στρατηγική για τις ε, μεταφορές που να μας λέει πώς μπορούν να συνδυαστούν οι μορφές μεταφορών, δηλαδή ε, οδικές, οδομικές κτλ. Αυτό χρειάστηκε χρόνο για να το κάνουν, αλλά είχε έννοια γιατί κατόπιν όλες οι επενδύσεις εντάσσονταν σε μία λογική. Αυτό κράτησε βέβαια πολύ σε κάποιες χώρες. Αυτό σήμαινε ότι απελευθερώθηκαν και οι πόροι αργότερα. Αλλά νομίζω πως είχε έννοια. Και στο μέλλον θα αξιοποιήσουμε παρόμοιες στρατηγικές. Σας παρακαλώ, υποστηρίξτε μας να αποφύγουμε το 1 3 αποφασίστε όσο ταχύτερα γίνεται το πολιτές πλαίσιο όσο ταχύτερα το αποφασίσουμε τόσο ταχύτερα θα το εφαρμόσουμε για τους ίδιους πόρους και την απάτη του ΦΠΑ Νομίζω ότι έχει υπάρξει ουσιώδης πρόοδος. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από πολύ επιμελή ανάλυση με τη συμμετοχή της Όλαφ και άλλων ε, υπηρεσιών θεωρούμε ότι προκύπτουν 2,8 δις ε, απώλειες από απάτες. Τα συζητήσαμε και με τις Βρετανικές Τελωνιακές Αρχές και νομίζω ότι έχει υπάρξει βελτίωση. και σε άλλους τομείς. Έχει υπάρξει βελτίωση. Γιατί θεωρούμε ότι τώρα έχουν πέσει στα δύο δις οι απάτες. Αυτά που αναφέρατε για το 95, δεν ξέρω. ΦΠΑ λέει πρόεδρος. Τι πράγμα? Για το ΦΠΑ. Ναι, ναι, άλλο τα τελωνία, άλλο το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθω. Αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα δικό μας. Υπάρχουν διάφορες ε, προσπάθειες για να το επιλύσουμε. Πριν από μερικέ μέρες συζήτησα με εκπροσώπου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μου είπαν ότι είναι υπό εξέλιξη μια προσπάθεια Ας πούμε, εάν μια επιχείρηση θέλει να παραδώσει εμπορεύματα από τη Βαβαρία στην Ελλάδα, θα πρέπει να ε, διασφαλίζει ότι θα γίνεται σωστά η πληρωμή του ΦΠΑ στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να γίνει. Δεν λειτουργεί στην πράξη, άρα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τώρα το κόστος για τις ιδιωτικές πτήσεις, ε, ότι αυξάνεται τώρα δεν τα ξέρω απ' έξω, αλλά έχουμε μια σύμβαση πλαίσιο για, αυτή την, ε, για αυτές τις πτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δαπανίσουμε όσα προβλέπεται στη σύμβαση πλαίσιο, αλλά πρέπει να υπάρχει μια προκήρυξη, ούτως ώστε αν χρειαστούμε ένα αεροπλάνο ε, ιδιωτικό. Έχουμε λοιπόν ήδη ένα συμβόλαιο που μας λέει από ποια εταιρεία θα τον νοικιάσουμε. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πάντα ελέγχεται πάρα πολύ ε, αν οι τιμές που μας δίνουν αυτές οι εταιρείες σε σχέση με τις ε, κανονικές πτήσεις. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Τώρα το θέμα του κράτους δικαίου. Αυτά που οι υποθέσεις που βλέπουμε στην Τσεχία. Κοιτάξτε. Εντάξει, υπήρξαν κάποια θέματα δημοσίευσης, αλλά η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη δεν μπορώ να τοποθετηθώ εδώ επί της ουσίας. Πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με κανόνες συμμόρφωσης και με το κράτος δικαίου. Και αν εμείς ως θεσμοί καλούμε να γίνονται αυτά σεβαστά, πρέπει και εμείς ε, να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο τήρηση αυτών των κανόνων. Οπότε παρακαλώ να κατανοήσετε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να εκφραστώ επί της ουσίας γιατί θα ήταν αντίθετο με τους κανόνες. Τι έχουμε κάνει. Ως Επιτροπή καταρτήσαμε μια τελική έκθεση η οποία απεστάλλει πρώτα απ' όλα στην τσεχική πλευρά για να τοποθετηθεί επ' αυτής. Και υποθέτω ότι όσο δεν έχουμε λάβει την τοποθέτησή τους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα ολοκληρωθεί όταν με βάση τη γνωμοδότηση και των ενδεχομένων συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών η Επιτροπή θα κάνει την εντελώς τελειωτική έκθεση με τα πορίσματα. Υποθέτω ότι θα γίνουν όλα αυτά κατά τα μέσα ή κατά το δεύτερο ήμιση του 2020. Και τότε θα το συζητήσουμε δημοσίω. Με, με συγχωρείτε, ε, με συγχωρείτε. Εντάξει, μπορεί να μην σα αρέσουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, βέβαια όλα αυτά δεν, δεν μα διασκεδάζουν όταν τα διαβάζουμε σε εφημερίδε. Κοιτάξτε, ε, τηρείτε η εμπιστευτικότητα. Με συγχωρείτε, εμένα δεν με διασκεδάζουν αυτά. Δεν γελάω. Εγώ τηρώ τους κανόνες ε, του παιχνιδιού. Ό,τι κάνετε εσείς είναι δικό σας θέμα. Εγώ πρέπει να τηρήσω τους κανόνες. Δεν μπορώ να αποκλίνω ούτε ελάχιστα. Τώρα αυτή η αρπαγή υγεών. Και εμείς εκπλαγήκαμε όταν είδαμε ότι στην Σλοβακία το το μητρό, το κτηματολόγιο. Δεν τα πάει τόσο καλά, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και από την ελληνική πείρα ξέρω ότι αυτά δεν διορθώνονται από τη μία χρονιά στην άλλη, αλλά έχουμε συνέστηση του προβλήματος και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιλύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να κάνω μια παρατήρηση, αγαπητέ Επίτροπε γιατί θα παρατηρήσατε ότι δημιουργήθηκε και μια αναταραχή εδώ στην αίθουσα. Όταν διαρρέει στη δημοσιότητα μια τέτοια έκθεση, καταλαβαίνετε ότι αυτό αλλάζει και τους όρους του παιχνιδιού. Γιατί θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορούμε και εμείς εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Όταν αδημοσίευτες εκθέσεις έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Αυτό δυσκολεύει και το δικό μας έργο και το δικό σας έργο, γιατί ε, έχουμε λάβει όλη γνώση πλέον ε, των στοιχείων που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Ταυτόχρονα όμως ο Επίτροπος δεν δύναται, δεν δικαιούται να λάβει θέση γιατί δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τους όρους του παιχνιδιού, με τους κανόνες. Και ο, η Επιτροπή Προπολογισμών ε, μάλιστα αποφάσισε χθες να ε, απευθυνθεί στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και να ε, ρωτήσει πώς ακριβώς πρέπει να χειριστούμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δώσω το λόγο στους Σκιώδης, η κυρία ε, Διαδικαστικό. Συγγνώμη. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο. Έχουμε περάσει μία ώρα και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να υποβάλουμε ερωτήσεις προς εσάς, πέρα από την εισηγήτρια. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο. Θέλω να εξασφαλίσετε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να ε, υποβάλουμε τις ερωτήσεις μας. Αλλά με ισοτιμία μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Γιατί έχει πέρασει μία ώρα και δεν έχουμε καταφέρει να υποβάλουμε ούτε ένα ερώτημα ακόμη. Πρόεδρος, ναι, έδωσα 20 λεπτά στο ελεγκτικό συνέδριο, 10 λεπτά στον Επίτροπο και προφανώς ε, πρέπει οι φορεί και τα όργανα που εκπροσωπούν να έχουν τη δυνατότητα ε, να, να τοποθετηθούν. Ε, λοιπόν, δίνω το λόγο στη συνάδελφο Πένκοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου που παρουσίασαν την έκθεσή τους. Ευχαριστούμε και τον, ευχαριστώ και τον Επιτροπο Χάν που βρίσκεται εδώ και απαντά στις ερωτήσεις μας. Έχουμε λάβει κάποιες απαντήσεις και γραπτός. Ε, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα θα σας τα πω. Θέλω να ρωτήσω, ε, να υποβάλω ένα διευκρινιστικό ερώτημα. Σε μία από τις ε, ερωτήσεις που σας αποστήλαμε, θέλουμε να, θέλω να κάνω ένα βηματάκι πίσω. Ξέρω ότι συζητούμε κυρίως για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Θέλω όμως να σας θέσω ένα ερώτημα για την τρέχουσα περίοδο. Ακούσαμε τα στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά απορρόφησης και επιλογής ε, υπό το τρέχον πι δέλτα πι και την κοινή διαχείριση. Το ερώτημα μου είναι ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν αφορούν τα ταμεία συνοχής. Μπορούμε να λάβουμε όμως στοιχεία ε, για τα ποσοστά απορρόφησης όλων των προγραμμάτων που εντάσσονται στο ΠΔΠ. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να μην έχετε την απάντηση αυτή τη στιγμή για να μας τη δώσετε. Όμως αν έχει δημοσιευτεί μια τέτοια πληροφορία ε, θα σας παρακαλούσα κύριε Πίτροπε να μας την αποστείλετε γραπτός. Ο κύριος ε, Σωστέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλές εντάσεις στην Επιτροπή σα σήμερα, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να επιστρέψω σε κάποια στοιχεία, κυρίως των γραπτών απαντήσεων που στείλατε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα καταρχάς να συνεχίσω με αυτό που έλεγε η Πρόεδρος για την απάτη ΦΠΑ, που είναι τεράστια. Ε, και βρεθήκαμε να διαπραγματευόμαστε νύχτες ολόκληρες ε, για να έχουμε ένα συγκεκριμένο προπολογισμό, το να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό απάτης ΦΠΑ είναι πραγματικά απογοητευτικό, δυσάρεστο και πέραν ε, του συναλλικού ποσοστού απάτης ΦΠΑ θα ήθελα να γνωρίζω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει να δώσει συγκεκριμένες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για θέματα ΦΠΑ, κυρίως για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα ε, η ηλεκτρονική ε, απάτη ΦΠΑ, μάλλον η απάτη ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό ε, εμπόριο είναι περί ήδη 500 δις ευρώ ετησίως, 5, συγγνώμη, 5 δις ευρώ ετησίως ε, και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στοιχεία θα πρέπει να μα ανησυχούν περισσότερο τι γίνεται με αυτή την απάτη ΦΠΑ. Θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό που ανέφερε ήδη η Πρόεδρος για θέματα Απάτη ΦΠΑ. Δεύτερον, το 2018 μπορέσαμε να παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα έχει ένα νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και θα ήθελα να ξέρω βάσει ποιων στοιχείων του προηγούμενου πλαισίου έγιναν συγκεκριμένε προτάσεις. Και θα ήθελα επίσης να μου πει ο Επίτροπο ε, τι άποψη έχει για μια πιο σύντομη περίοδο προγραμματισμού που θα επιτρέπει να ε, ευθυγραμμίζεται και με την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Τρίτον, κάτι που αναφέρεται συχνά στις απαντήσεις σας, τα ποσοστά σφαλμάτων και τη μεθοδολογία. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον προβλέπετε να πάρετε λέα μέτρα για να απλοποιήσετε αυτά τα ποσοστά ασφάλματος, να εναρμονίσετε τις μεθοδολογίες και να φροντίσετε ο καθένας να χρησιμοποιεί το ίδιο ποσοστό σφάλματος, γιατί αυτοί που ξέρουν να τα αξιολογήσουν μπορούν να δούνε πώς ε, θα βελτιώσουν τα πράγματα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε δηλαδή τη συλλογή δεδομένων, κυρίω για τα θέματα τα οποία μοιραζόμαστε μεταξύ των κρατών μελών και ε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Επίσης, για τις απαντήσεις σας ε, στις ερωτήσεις 34 και 35, στις οποίες επιμένετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα διευκρινίσει τα θέματα του καταμερισμού του σε επόμενης προγραμματικής περίοδου για το στρατηγικό προγραμματισμό για την επόμενη γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκοπεύει λοιπόν να συμπεριλάβει λίγο καλύτερα τις πτυχές που αφορούν τις επιδόσεις ως βάση για τον επόμενο πολιετής ε, κύκλο στρατηγικού προγραμματισμού και να μας πει ε, τι διαφορετικό προβλέπει να κάνει όσον αφορά τα νέα προγράμματα ε, σε σχέση με αυτά που είχαμε στον προηγούμενο κύκλο. Κύριε Κάμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Επειδή ήσασταν και Επίτροπος ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και επειδή είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα, θέλω να ξανατονίσω ότι δεδομένης της επιφυλακτικότητας που συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια όσον αφορά τις υψηλές, τις υψηλές δαπάνες για διαρθρωτικά ταμεία και γεωργικά ταμεία, είναι προφανές ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν αποκαλύπτεται μια τέτοια υπόθεση στην Τσεχία, ελέγχεται από εσάς, ελέγχεται από τον Όλαφ και καταλήγει ε, στο συμπέρασμα κανείς ότι προφανώς για όλα αυτά θα έπρεπε η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να είχε ενημερωθεί έγκαιρα. Και το διαπιστώσαμε χθες το βράδυ. Όλοι μας οι φόβοι τελικά επιβεβαιώθηκαν. Μάλιστα είχατε αποστείλει και συγκεκριμένη γνωμοδότηση προς την τσεχική κυβέρνηση. Και τώρα μας λέτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλους έξι μήνες όταν πια θα έχουν Ολοκληρωθεί και οι διαπραγματεύσει για το νέο πι όχι, ο ρόλος μας είναι διαφορετικός. Και εγώ ως βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, έχω διαφορετικό ρόλο. Ή έτσι τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι εγώ. Όταν με τα δικά μας χρήματα ενισχύονται ολιγαρχικές δομές, σε όποια χώρα και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το πρόβλημα είναι πραγματικό, είναι υπαρκτό και είναι σοβαρό. Διότι ο Μπάμπης δεν έχει μόνο την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ε, στην Τσεχία έχει είναι ο μεγαλύτερος εργοδότη και στη Βιτεμβέρχη. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος ακινήτων και στην Ανατολική Γερμανία. Σε πολλές περιοχές και σε πολλές πόλεις. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε μέσω τη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όταν υπάρχει απάτη, στην οποία περιλαμβάνονται ευρωπαϊκά κονδύλια, στα οποία έχει υπάρξει κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα πρέπει εδώ εμεί να το συζητάμε. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Ολομέλεια. Με όλα τα στοιχεία ανοιχτά και στο τραπέζι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τις απαντήσεις που λάβαμε σε ερωτήσεις μας σχετικά με την υπόθεση Μπάμπης πρέπει να τις λαμβάνουμε έγκαιρα και γρήγορα. Πολλές φορές καθόμαστε και ψηρίζουμε πολύ μικρότερα ποσά σε διάφορους προϋπολογισμούς, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε υποθέσεις, υποθέσεις στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχία, όπου υπάρχουν, υπάρχει κατάχραση τεράστιων ποσών και περνάει περνάνε τεράστια χρονικά διαστήματα έω ότου αποκτήσουμε τη δυνατότητα τελικά να συζητήσουμε τις υποθέσεις αυτές. Αυτό το θέμα θα πρέπει να δημιουργήσει συγκεκριμένες επιπτώσεις και για τα πολιτικά πράγματα στην Τσεχία. Όταν, έχει μια, όταν υπάρχει μια τέτοια υπόθεση, προφανώς και θα πρέπει να επιβάλλονται επιπτώσεις. Και το ζήτημα εδώ είναι ποια είναι η στάση της κοινή γνώμης τη της Έχετε δει ότι έχουν γίνει διαδηλώσεις με 300.000 ανθρώπους στους δρόμους. Αυτή η αριθμή δεν είναι μικρή για την Τσεχία. Επομένως, προφανώ πρέπει σε αυτή τη δυναμική και εμεί να ασκήσουμε ποιήση. Γι' αυτό σα καλώ δημοσιεύστε όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να γίνει ανοιχτή συζήτηση. Προσπαθήστε κι εσείς στα δικά σα θεσμικά όργανα να αποφύγετε την απάτη, ώστε στο μέλλον να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιες υποθέσεις. Ωραία. Πρόεδρος. Βλέπετε ότι η ατμόσφαιρα εντός της Επιτροπής μας δεν είναι η καλύτερη Δυστυχώς η έκθεση διέρευσε. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε πλέον. Εγώ θα απευθυνθώ και στην νομική υπηρεσία για να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να λάβουμε εμείς αυτή την οριστική έκθεση. Ο κύριος ε, Κρούς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω, κύριε Χάν. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της διαλειτουργικότητας Είναι πολύ σημαντικό το, το ζήτημα αυτό. Και ε, είπατε ότι υποστηρίζετε και τους απλούς κανόνες. Κάτι το οποίο βεβαίως είναι προφανές. Η διαλειτουργικότητα μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον υπάρχουν απλοί και κοινοί κανόνες. Σας ερωτώ λοιπόν. Αυτή η διακήρυξη δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι πρώτα και κύρια η Κομισιόν που είναι εκείνη που λαμβάνει την πρωτοβουλία για τη θέσπιση νέων κανόνων ε, να δεσμεύεται από μια τέτοια ε, από μια τέτοια αρχή. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση ε, όσον αφορά την απλοποίηση των κανόνων, τη θέσπιση νέων απλών αποτελεσματικών κανόνων. Αντίστοιχε συστάσει άλλωστε έχει υποβάλει και το ελεγκτικό συνέδριο. Η κυρία Λίνστρον μα είπε ότι η περιπλοκότητα των, δομή ε, της δομής των προϋπολογισμών και των διαδικασιών χρηματοδότησης είναι πρόβλημα. Οπότε σας καλούμε εμείς, πρώτα και κύρια εσείς, να τεθείτε επικεφαλής αυτή τη διαδικασία απλοποίηση των, των κανόνων και εμεί θα σα υποστηρίξουμε. πρόεδρο. Κύριο Χάν και μετά θα ακούσουμε άλλους τέσσερις ευρωβουλευτές. Για το πρώτο ερώτημα. Ναι, μπορούμε να σας δώσουμε τα στοιχεία όσον αφορά τα, τα ποσοστά απορρόφησης των διαφόρων προγραμμάτων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σχετικά με, την, ε, με το ζήτημα του, του, του ΦΠΑ. Εγώ θα πρότεινα να το συζητήσουμε σε ξεχωριστή, με ξεχωριστή αφορμή αυτό το θέμα, σε ξεχωριστή συνεδρίαση όπου θα μπορούν να έχουμε εστίαση και σε ζητήματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαλειτουργικότητα. Εγώ ξέρετε ότι θέλω να ενισχύσω την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να ενισχυθεί και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. Σας το λέω ανοιχτά. Υπάρχουν μια σειρά από κράτη-μέλη, τα οποία έχουν εκφράσει σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς μια τέτοια προοπτική με διάφορα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Δεν θα σας τα αναφέρω τώρα όλα. Απλώς για εσάς αυτό που είναι σημαντικό ε, είναι, θα ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να με υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη προς μια τέτοια κατεύθυνση της ενίσχυσης ανταλλαγής δεδομένων και προφοριών. Και με αυτό να απαντήσω και στον κύριο Γκρού. Για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε προτείνει 80 απλοποιήσεις σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες και αυτό σημαίνει στην πράξη ότι θα υπάρξει μείωση του ποσοστού σφάλματος. Το ουσιώδες όμως, και το είπα και εισηγητικά, είναι ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Την προηγούμενη φορά έγιναν 73 τριμερείς διάλογοι και για να είμαι ειλικρινής δεν βοήθησε και πολύ η διαδικασία αυτή στην απλοποίηση. Και, έπειτα υπάρχει στα κράτη-μέλη και η διαδικασία του gold plating, της, ε, του κανονιστικού υπερθεματισμού, που σημαίνει ότι ε, έρχονται τα κράτη-μέλη και επιβάλλουν νέους κανόνες, εξειδικευμέν, πιο εξειδικευμένους κανόνες, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι τελικοί δικαιούχοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεωργοί, να μην απευθύνονται ε, στα ευρωπαϊκά προγράμματα για χρηματοδότηση, γιατί οι κανόνες είναι υπερβολικά επαχθείς και δεν μπορούν να τους στηρίσουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα να σας καλέσω να μας υποστηρίξετε, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τη διαλειτουργικότητα. Όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος και τις διαφορετικές μεθοδολογίε που χρησιμοποιούνται, ε, το θέμα, ξέρετε, έχει, έχει συζητηθεί τόσο πολλέ φορέ. ε, που νομίζω ότι εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Το ελληνικό συνέδριο έχει βεβαίως τη δική της οπτική. Εμείς από πλευράς Κομισιών και κρατών μελών ελέγχουμε όλες τις συναλλαγέ, τα κράτη-μέλη δηλαδή είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν όλες τις συναλλαγές που γίνονται. Το ελεγκτικό συνέδριο βεβαίως λόγω του ετήσιου χαρακτήρα της υποβολής των εκθέσεων εξετάζει τις συναλλαγές με μια διαφορετική, από μια διαφορετική σκοπιά, γι' αυτό και δημιουργούνται διαφορετικά ποσοστά ασφάλματος. Τελική παρατήρηση για τα όσα είπε η συνάδελφος των Πρασίνων και για σένα Μόνικα. Νομίζω ότι και ο όρος τελική έκθεση είναι κάπως παραπλανητικός, διότι πρόκειται για μια προκαταρκτική διαπίστωση εσωτερική της Κομισιόν, με την οποία καλούμε την άλλη πλευρά να τοποθετηθεί. Και στη βάση των συζητήσεων που θα γίνουν, έτσι προβλέπουν οι κανόνες του κράτους δικαίου, θα υπάρξει στο τέλος η πραγματική τελική έκθεση, αν θέλετε. Εγώ δεν μπορώ να καθορίσω τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ όμως, επαναλαμβάνω ότι είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω τους κανόνες του ισχύοντε. Αν εσείς επιθυμείτε να του αλλάξετε τους κανόνες αυτούς. Εγώ ευχαρίστως να τηρήσω πλέον τους νέους κανόνες που θα θεσπίσετε. Αλλά μην με κατηγορείτε για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ε, τηρώ τους κανόνες που ισχύουν και που με δεσμεύουν. Δεν δημοσίευσα δυστυχώς εγώ ε, την έκθεση αυτή, δεν είναι δική μου ευθύνη. Με κάποιον τρόπο τελικά διέρευσε η έκθεση αυτή. Προφανώς και είναι πολύ δυσάρεστο το φαινόμενο αυτό. Μπορείτε να το συζητήσετε, εγώ δεν μπορώ να σας επιβάλλω τι θα συζητήσετε και τι όχι, αλλά και στην Ολομέλεια μπορείτε να το συζητήσετε δηλαδή, αλλά εγώ καταλαβαίνετε ότι έχω, είμαι υποχρεωμένο να τηρήσω του κανόνε και επομένω όσε ερωτήσει και αν μου θέσετε αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Κύριε Τσιντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε δίκιο πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση κάποιοι μεν τηρούν τους κανόνες και άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Εγώ ως επιχειρηματίας δεν έλαβα καμία ευρωπαϊκή ενίσχυση και από σφάλμα ε, βρέθηκα εδώ να ασχολούμαι με το ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα. Ποτέ δεν είδα τόσα ασφάλματα, τόσα λάθη, τέτοια πράγματα ε, φρικαλέα, πράγματα τα οποία δεν είχαν κανένα νόημα και έπρεπε να τα παρουσιάσουμε. Μετά από μερικά χρόνια έγινε ένας νέος έλεγχος και παρά το γεγονός ότι είχα κάνει 10 φορές, ε, βρέθηκα τελικά να παρουσιάζω τα ίδια έγγραφα 100 φορές. Ένα παράλογο πράγμα. Εγώ ήμουν ένας μικροεπιχειρηματίας εννοείται κύκλο εργασιών 10 εκατομμύριων, τίποτα το ενδιαφέρον. Πείτε τώρα εσείς ένα μικρό επιχειρηματία ότι ε, υπάρχει απάτη τέτοιου μεγέθους. Εδώ εκατο... μιλάμε για δισεκατομμύρια ενισχύσεις. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποφασίσουμε ότι για το νέο πρόγραμμα και τη νέα προγραμματική περίοδος από το 2000 21 στο 2027 θα ε, αποφασίζεται σε ποιον θα ανατίθεται αυτά τα κονδύλια. Θα χρειαστούμε τρία χρόνια για κάτι τέτοιο. Ε, κάνετε λάθος ως προς το εξής κύριο Πίτροπε. Αυτή δεν είναι μια τελική έκθεση. Εγώ συζητούσα τρία χρόνια με το θέμα ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκθεση που ήρθε για την ε, Τσεχία είναι τελική έκθεση στην οποία διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι τελική, οριστική, υπό την έννοια ότι ακόμα θα υπάρξει και έλεγχος όσον αφορά τους περιορισμούς που θα προκύψουν. Αλλά το ότι υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων, αυτό δεν είναι πλέον θέμα προς συζήτηση. Και ε, έχω και άλλες ερωτήσεις και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται και με το χρονοδιάγραμμα θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε. Επίσης θα ήθελα να ξέρω διότι στη Σλοβοκία είχαμε περιπτώσεις απάτης με ευρωπαϊκές ε, επιδοτήσεις ε, και επιλήθηκαν. Ξέρετε πόσες φορές χρειάστηκε να χρεοκοπήσουν γεωργοί επειδή έπρεπε να επιστρέψουν ή τελικά τους κοβόταν η επιδότηση και τελικά βρεσκόντουσαν χρεοκοπημένοι. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνετε ενώπιον των κρατών μελών. Πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να προστατευτούν από αυτά τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα εφαρμόσετε τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων στο μέλλον. Αν ένας πολυεκατομμυριούχος έχει επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται σε ενισχύσεις με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, σε γεωργικά ζητήματα, πώς ε, θα μπορέσει, για παράδειγμα, να μετεγκατασταθεί αλλού και να λάβει πάλι ευρωπαϊκή ενίσχυση. Θεωρώ ότι πηγαίνουμε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Και επίσης, θα ήθελα να ξέρω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην επανεληφθούν τέτοια πράγματα. Και αυτή είναι η γενική ερώτηση επί τη οποία πρέπει να απαντήσουμε σήμερα. Κάτι ακόμα. Όταν βλέπουμε πώς τα κράτη-μέλη βρίσκονται συνεχώς ε, ενώπιον των δικαστηρίων, ε, θα ήθελα να ξέρω μήπως ε, ελοχεύει ένας κίνδυνος, μήπως υπάρχει κίνδυνος κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, υπάρχει διαφθορά και σύγκρουση συμφορώντων, μήπως πρέπει να αλλάξει το σύστημα ελέγχου τελικά. Διότι σήμερα συζητάμε τα θέματα του Αντρέι Μπάμπιτς. τα είπαμε γενικά γιατί υπάρχουν και οι περίπτωση της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορούμε να στήσουμε ένα σύστημα το οποίο είναι πραγματικά αποτελεσματικό για τους ελέγχους ε, για αυτές τις ε, δημόσιες ενισχύσεις. Ευχαριστώ, η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. να ευχαριστήσω τους ε, ελεγκτές της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Λαζάρου και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Χάν που βρίσκεται εδώ σήμερα για πρώτη φορά με τη νέα του ιδιότητα ως Επίτροπος Αρμόδιος για το προπολογισμό. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ξέρω την αποφασιστικότητά σας και την αφοσίασή σας και είμαι βέβαιη ότι θα αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που έχετε ενώπιόν σας. Καταρχάς για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως είδαμε, είχαμε ε, απόφαση το 17 Δεκεμβρίου του 2013. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με τη περίοδο του 2014-2020. Είχε καθυστερήσει να υποβληθεί το σχέδιο κειμένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ομάδα του Μπαρόσο. Τώρα όχι γιατί εγώ ήμουν επίτροπος τη ε, της ομάδας του Γιούνκερ, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε ενώπιον ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την πρόταση του πολιετίου πλαισίου για το 2021, 2021, 2027 από τις 2 Μαΐου του 2018. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορεί να απεμπλακεί η κατάσταση στο Συμβούλιο. Το συζητήσαμε για παράδειγμα στην Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη και κοιτάμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και διάθεση από πλευρά Συμβουλίου. Γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Δεν ε, με ικανοποιεί καθόλου να βλέπω ότι δεν προχωρά το πολιετές ε, και θα είναι σχεδόν αδύματο να ξεκινήσει η εφαρμογή της ε, νέας προγραμματικής ε, περίοδου από 1η Πρώτου του 2021. Αυτό σημαίνει ότι ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να υπάρχει πρόβλημα για πάνω από 100.000 προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και για να ξεκινήσουν και τα νέα προγράμματα της προγραμματικής περίοδου. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο για να απεμπλακεί λοιπόν αυτή η κατάσταση και να υπάρχει πρόοδος στο συντομότερο δυνατόν. Έγιναν μόνο τρει τριμερείς διάλογοι και την προηγούμενη φορά κάναμε 173 τριμερεί διαλόγου για να αποφασιστεί το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω και την ευθύνη των κρατών μελών. Θεωρώ ότι εμεί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφεύγουμε να συζητούμε αυτή την κατάσταση. Σε όλε τι εκθέσει ε, που έχουμε, Φαίνεται ότι το 90% των σφαλμάτων και των περιπτώσεων απάτης θα μπορούσαν να είχαν διαπιστωθεί αν είχε γίνει ο έλεγχος καταλήλως στο πρώτο επίπεδο ελέγχου. Αυτό σίγουρα είναι πρόβλημα και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την απλοποίηση. Όπως ξέρει πάρα πολύ καλά ο Επίτροπος Χάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια ριζοσπαστική απλοποίηση και είμαι βέβαιη ότι θα τον υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πολλά κράτη-μέλη προτιμούν να έχουν όλη αυτή την επιπλέον επιβολή κανόνων. Υπερβολική νομοθεσία και επιπλέον κανόνε. Και θα ήθελα να ξέρω και τι θα γίνει και με τον προπολογισμό. Η Ιζαμπέλ Γκαρθία Μουνιό τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση του διεθνούς, ε, της Διεθνούς ε, Ομάδας Διαχείρισης, της IMG. Βλέποντας τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το ερωτηματολόγιο για την απαλλαγή του 2018, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, με τελεσίδικη απόφαση 31 Ιανουαρίου για την περίπτωση του AMG. Και είναι σαφής η απόφαση, καταδικάζει τις δύο αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του AMG για ε, όσα έγιναν βάσει μιας έκθεσης της Όλαφ στην οποία βάσει της ε, δικαστικής απόφασης ε, τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν ήταν παραβίαση του δικαίου και σε διεθνές ε, λογιστικό επίπεδο και όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρεται στη στάση του IMG. Θα πρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι και να τηρήσει τα όσα προβλέπει η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να α, ε, τηρήσει τα της απόφασης ζητάει από τον IMG να αποδείξει ότι όντως έχει καθεστώς διεθνούς οργανισμού όταν αναγνωρίζεται ως τέτοιο εδώ και 20 χρόνια. Επίτροπε Χάν, πέραν από το γεγονός ότι θα ήθελα να σας πω να δείτε τις ε, παραγράφους 183 με 187 της εκθέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαλλαγή του 2018, θα ήθελα να σας θέσω και τις ίδιες ερωτήσεις που έκανα και στον πρώην ε, Επίτροπο Έτιγκερ τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, τηρεί μια τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάθονται σε ένα τραπέζι με την IMG για να βρουν επιτέλου μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Αυτό θα αποφύγει στη νέα προσφυγή στο δικαστήριο και την εξαφάνιση ενός οργανισμού με πάνω από 200 ε, υπαλλήλους που εδώ και 20 χρόνια εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποτελεσματικό ε, τρόπο και ε, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε στάση τόσο ριζικά ενώπιον αυτού του οργανισμού το 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος, ποιος έχει φύγει. Να κάνω και εγώ τότε την ερώτησή μου για την περαιτέρω εξέλιξη. της ε, υπόθεσης της Τσεχίας. Είναι η τελική έκθεση. Γιατί είχατε επαφές εδώ και πολλούς μήνες με την ε, Τσεχία Έχετε ακούσει τις απόψεις τους. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να τηρεί κανείς τους κανόνες. Αλλά θα πρέπει η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον και κλεισμένο των θυρών να συζητήσει τα θέματα αυτά. Καταλάβουμε τι τρέχει. Και να μην λάβουμε μέτρα μετά την απόφαση για το πολιτές πλαίσιο, αλλά πριν για διάφορα προγράμματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ακόμα 6 μήνες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, για το θέμα των κανόνων του παιχνιδιού, να κάνουμε μια συνεδρίαση και κλεισμένα των θυρών. Όχι δημόσια. Ω μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Να κάνουμε πιο αναλυτικέ ερωτήσει για τα θέματα συνοχής, γεωργίας και παρακαλώ έχετε το λόγο τώρα γιατί ακριβώς ε, μίλησα μέχρι να έρθετε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Με ενδιαφέρει τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Να κάνω μία ερώτηση για τις εκθέσεις αυτές. Οι οποίες, για την έκθεση αυτή για την Τσεχία η έκθεση αυτή αποδεικνύει σαφώς ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση του κυρίου Μπάμπης. Αυτό σημαίνει ότι η Τσεχία πρέπει να επιστρέψει τα ποσά αυτά. Αλλά εξακολουθεί ο κύριος Μπάμπης να είναι σε κατάσταση σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί είναι πρωθυπουργό. μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μπορεί λοιπόν ε, να θέσει βέτο για την έγκριση ε, του προπολογισμού ή του πολιετούς πλαισίου άρα αξιοποιεί αυτή τη θέση για τις επιχειρήσεις του. Μεγάλος κίνδυνος λοιπόν για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Και μπορεί να προκύψουν και περαιτέρω ζημίες, πολύ μεγαλύτερες. Δεν θα ήθελα λοιπόν να είναι υπεύθυνη η Τσεχία για αυτή τη συμπεριφορά. Και τελικά να πληρώσουν οι Τσέχοι φορολογούμενοι τα σπασμένα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μεγάλα ποσά. Και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το δεύτερο εξάμενο του 2020. Μα δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τόσο πολύ. Τι είναι αυτή η καθυστέρηση. Νομίζω ότι το πνεύμα των συνθήκων σημαίνει ότι πρέπει να δράσει επιτέλου η Κομισιόν για να αποφευθούν περαιτέρω ζημίες. Ευχαριστώ πολύ. Η Κατερίνα Κινίτσι και μετά θα ολοκληρώσουμε. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο και καλή δουλειά να σας ευχηθώ και να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους του Ελεκτικού Δικαστηρίου. Ε, Ταμείο Συνοχής, ε, το ακούσαμε συνεχώς, ε, σφάλματα και απάτη. Ακούσαμε το ελεγκτικό συνέδριο και ακούσαμε και εσά κύριε Επίτροπε και ακούσαμε ότι κάνατε και δύο αναφορά στην Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην οποία εμπιστευόμαστε όλοι. Επομένως θα ήθελα και εγώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορέσει να γεννηθεί επιτέλους ε, με όλους τους πόρους που χρειάζονται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της. Η παρέμβαση της Όλαφ ε, και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, έχουν στόχο να αναδειχθούν τα σφάλματα και οι παρατυπίες και η απάτη. Αλλά όπως είπε και προηγουμένως η ε, πρόεδρος Χολμάγερ, η, πρέπει να προλάβουμε τις καταστάσεις. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει απλοποίηση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα αρκέσουν αυτά. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να προλάβουμε σφάλματα και απάτη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για σήμερα, διότι δέχομαι ευχαρίστως την πρόταση της Προέδρου να το συζητήσουμε και κλεισμένον. Οι συνάδελφοί μου εδώ μου είχαν ήδη κάνει αυτή την πρόταση. Μου το ψιθυρίζανε εδώ οι συνεργάτες μου. Βεβαίως, αλλά σας παρακαλώ, και κλεισμένον των θυρών σημαίνει και κλεισμένον των θυρών. Όχι κάποιοι να βγαίνουν από τις συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών και να κάνουν συνέντευξη τύπου Γι' αυτό παρά το ότι οι συνεργάτες μου εδώ μου λέγανε «Μα κάντε την πρόταση αυτή», εγώ δίσταζα. Σας παρακαλώ λοιπόν, θα πρέπει να είναι εμπιστευτική η συζήτηση. Και ό,τι λέμε εδώ μέσα θα πρέπει να σας βοηθούν αλλά να μην βγαίνετε και αμέσως όταν τα λέτε στον τύπο. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω βέβαια ότι έχετε μια πολιτική προσέγγιση στην οποία δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Και φυσικά θα σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν εκφράστηκε το δικαστήριο για το αν και κατά πόσο είναι διεθνής οργανισμός αυτό το IMG. Θα πρέπει να μας αποδείξει ότι έχει αυτό το καθεστώς για να έχουμε δυνατότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα μαζί τους. Τους στείλαμε μία επιστολή και τους ζητάμε να μας εξηγήσουν τι γίνεται. Τώρα εγώ δεν ξέρω. Εάν έγινε σωστά η εξέταση αυτής της ε, περίπτωσης. Αλλά πρέπει όπως και για κάθε άλλο θέμα να τηρούμε τους κανόνες όπως είναι. Αν αλλάξουν θα σεβαστούμε τους νέους. Αλλά τώρα πρέπει να σεβαστούμε αυτά που γίνονται. Όσον αφορά το ποσοστό σφαλμάτων, μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ με την απλούστευση στην ε, ε, πολιτική συνοχή. Ξέρετε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τελικούς δικαιούχους, είναι μικρές επιχειρήσεις, ε, ενώσεις κτλ. Και Όλοι αυτοί δεν μπορεί βέβαια να είναι οι δήμονες για τα ενωσιακά θέματα. Μπορεί λοιπόν να προκύψουν σφάλματα. Και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Πάνω από 99% των περιπτώσεων σφαλμάτων είναι απλώς σφάλματα, όχι απάτες. Είναι σφάλματα στην ερμηνεία κάποιων ε, κανόνων ε, για το τι μπορεί να λάβει ενισχύσεις και τι όχι. Και είναι σαφές όσο, όσο πιο περίπλοκοι είναι οι κανόνες τόσο πιο διαφορετικές μπορεί να είναι και οι ερμηνείες τους. Γι' αυτό αυτός, αυτή η προσέγγιση ενιαίου ελέγχου, το single audit approach, θα μας βοηθήσει να έχουμε απλούς κανόνες, ούτως ώστε όλες οι υπηρεσίες ε, ελέγχου να ελέγχουν με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες μεθόδους. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και για τη συνεργασία και για τα επιπλέον, τα επιμέρους θέματα κατά τη διάρκεια του σίγουρα θα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Πρόεδρος. Νομίζω ότι για τα θέματα του ξεπλήματος ε, χρήματος και της απάντησης του ΦΠΑ που λέτε ότι μπορεί να είναι έως και 95 δις θα πρέπει να πούμε πολύ περισσότερα. Και για την Τσεχία. Πολύ θετικό αυτό που είπατε, να το συζητήσουμε και κλεισμένο των θυρών, γιατί αν διαβάσουν οι συνάδελφοι την έκθεση θα καταλάβουν ότι πρέπει να εξάγουμε και συμπεράσματα για το μέλλον. Η κυρία Κρέτσου το διατύπωσε πολύ σωστά για τις, ε, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου. Και ο συνάδελφος Πέτσου είπε πολύ σωστά ότι όπως λέει και το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο των ελεκτών για να δούμε εάν οι εθνικές αρχές ελέγχου πραγματικά κάνουν το καθήκον τους όπως θα έπρεπε. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Σας ευχαριστώ όλους και τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικά χρόνο για να συζητήσουμε. Οπότε θα σας ξανακαλέσουμε. Κύριε Επίτροπε, εσάς ούτως ή άλλως θα σας καλούμε τακτικά. Δεν είναι μόνο υποχρέωση, αλλά και η επιθυμία μας. Και εσάς και την ομάδα σας. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία, στην οποία προσβλέπουμε. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο 12. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Πένκοβα ειδική έκθεση για τα συστήματα πληροφορικής, για τη στήριξη των ε, συνοριακών ελέγχων. Ή να κάνουμε ένα λεπτό διακοπή. Äh, λοιπόν. λοιπόν, να δώσουμε δυνατότητα στην Μπετίνα Γιάκοψεν να παρουσιάσει την ειδική έκθεση. Γιατί η συγκήτριά μας βιάζεται. Κύριε Γιάκοψεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτήν την ειδική έκθεση για τα ευρωπαϊκά πληροφορικά συστήματα για την υποστήριξη των διασυνοριακών ελέγχων, συνοριακών ελέγχων. Από τη δημιουργία της, η περιοχή Σέγγεν επιτρέπει στους ε, ταξιδιώτες να παίρνουν από τη μία χώρα στην άλλη χωρίς συνοριακούς ελέγχους. Περιλαμβάνει 26 χώρες συνολικά η περιοχή αυτή. Η κατάργηση των εσωτερικών συνολικών ελέγχων ενίσχυσε την ε, σημασία της ενίσχυσης των ε, ε, ελέγχων που γίνονται στα εξωτερικά σύνορα. Και για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί μια σειρά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν κοινοποιήσει, απολεσθέντα έγγραφα, κλαπέντα έγγραφα, θεωρήσεις, δακτυλικά αποτελέσματα, ε, ε, ε, δακτυλικά αποτυπώματα, τον άσυλο. Το PNR επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με, τους, με το πώς και ποιοι περνάνε τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Αφήξεις και αναχωρήσεις. Πάνω από 600 εκατομμύρια έχει επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργικά έξοδα 61,5 κατέτος ευρώ. Ποιο ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός ε, του ελέγχου που κάναμε, ποιες είναι τα, ποια είναι τα βασικά πληροφορικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια, για την υποστήριξη ε, του ελέγχου των ε, συνόρων. Υπάρχουν λοιπόν η, η εθνική διάσταση και η ευρωπαϊκή διάσταση και τα συστήματα που επιτρέπουν τον έλεγχο εκείνων που εισέρχονται στην περιοχή Σέγγεν. Ε, κάναμε συνεντεύξεις με ανθρώπους από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, τη Frontex και τον Λύσσα. Κάναμε επισκέψεις στη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία. Επίσης υποβάλαμε μια μελέτη σε συνοροφύλακες σε ολόκληρη την περιοχή Σέγγεν και ε, λάβαμε και αναλύσαμε 951 απαντήσεις. Στη βάση όλων αυτών συμπεραίνουμε ότι οι συνοροφύλακες χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο και βασίζονται όλο ένα και περισσότερο σε αυτά τα συστήματα κατά την διενέργεια των, ε, ελέγχων, των συνοριακών ελέγχων. Ωστόσο, κάποια δεδομένα ακόμη δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα συστήματα, ενώ άλλα δεδομένα είτε δεν είναι πλήρη είτε δεν εισάγονται έγκαιρα. Και αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα ορισμένων συνοριακών ελέγχων. Ποια είναι τα βασικά πορίσματα. Στον έλεγχό μας ε, εξετάσαμε αν τα πέντε αυτά κράτη-μέλη είχαν δημιουργήσει εθνικά συστήματα ε, όπως αυτά προβλέπονται από το, τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαπιστώσαμε ότι τα συστήματα αυτά έχουν καλό σχεδιασμό για την διευκόλυνση των συνολικών ελέγχων και ότι τα κράτη-μέλη γενικά ε, ανταποκρίνονται και συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά δεν είναι πάντοτε ίσα ως προς την αποτελεσματικότητά τους, γιατί κάποια κράτη-μέλη ε, δεν αξιοποιούν πλήρως τα, τα δεδομένα που διατίθενται σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Αυτό πολλές φορές ε, δημιουργεί καθυστερήσεις και προβλήματα στην ε, διαχείριση των ελέγχων, στην αποτελεσματικότητά τους τα ωφέλη που, που παράγονται από τα πληροφορικά εργαλεία γενικά εξαρτάται από την ικανότητα των χρηστών να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι τα αυτόνομα συστήματα, περιβάλλοντα, ε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ε, επαγγελματίες να εξασκηθούν, αν θέλετε, σε διάφορες περιπτώσεις, προτού τις αντιμετωπίσουν στην πράξη. Για κάποιο αγνοούμενο παιδί, για παράδειγμα, ή τον εντοπισμό κάποιου τρομοκράτη. Γι' αυτό το λόγο η πρώτη σύστασή μας είναι η Κομισιόν να δημιουργήσει ε, συγκεκριμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για το ΣΥΣ2 και το ΒΙΣ. Επίσης, οι ορισμένες καθυστερήσεις στην εφαρμογή πληροφορικών συστημάτων στο Eurosur και το PNR πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το PNR σχεδιάστηκε για να εντοπίζονται τρομοκρατικά και άλλα σοβαρά εγκλήματα. Η σύγκριση του PNR με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε βάση δεδομένων όπως το SIS-2 επιτρέπουν στις αρχές να εντοπίζουν επικίνδυνους, ε, με μονομένα επικίνδυνα μεμονωμένα ε, άτομα. Το γεγονός ότι το PNR δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα πλήρως και η συγκρισιμότητα με τις βάσεις δεδομένων πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα ως προς τον εντοπισμό επικίνδυνων ατόμων. Το σύστημα ε, αξιολόγησης Schengen διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Υπάρχουν όμως, ε, υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων προθεσμιών για την ε, υποβολή εκθέσεων και για την εφαρμογή των ε, διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται. Στην πράξη λοιπόν μπορεί να περάσουν έως και δύο χρόνια έως ότου ε, κάποιο κράτος μέλος της Σέγγεν αρχίζει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των ε, σχεδίων δράσης του και ακόμα περισσότερα χρόνια έως ότου ε, ληφθούν τα πρώτα διορθωτικά μέτρα. Γι' αυτό η Κομισιόν θα πρέπει να επιταχύνει την ανέρεση και την αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Κατά τη διέλευση συνόρων, οι συνοροφύλακε χρειάζονται τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα άτομα που περνούν τα σύνορα και να επαληθεύσουν ότι πράγματι έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην Ένωση. Για παράδειγμα, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι γίνονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κοινοποίηση, αν υπάρχει ειδοποίηση ή αν υπάρχει πρόβλημα με το ταξιδιωτικό του έγγραφο. Οι περισσότερε ειδοποίησει. Ε, αφορούν απολυσθέντα έγγραφα ή κλαπέντα έγγραφα. Όταν υπάρχει λοιπόν μια αντιστοιχία ανάμεσα στη βάση δεδομένων που υπάρχει κεντρικά και στην βάση δεδομένων που τηρείται στο σημείο διέλευση συνόρων, τότε υπάρχει hit. Όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, ο αριθμό των hits σχεδόν τριπλασιάστηκε. Και ο τριπλασιασμός αυτός συμβαδίζει με τις ειδοποιήσεις που εισήχθησαν ε, τα τελευταία χρόνια, από 25 σε 75 περίπου εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο αριθμός αναζητήσεων στο σύστημα ε, αυξάνεται διαρκώς. Οι εθνικές αρχές, τις οποίες επισκεφτήκαμε στον έλεγχό μας, μας είπαν ότι ελέγχουν κάθε άτομο που προσπαθεί να διέλθει από τα εξωτερικά συνέδρια. Ωστόσο, στην έρευνα που διεξήγαμε στους συνοριοφυλάκες στις χώρες ε, Σέγγεν μας έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Οι, απο... απαντήσεις δείχνουν ότι πάνω από μη... οι μισοί συνοροφύλακες ομολόγησαν ότι πάνω από, πάνω από μία φορά ο καθένας κλήθηκε να αποφασίσει αν θα πρέπει κάποιος να περάσει τα σύνορα ε, ή όχι. Αυτό έχει σχέση με προβλήματα συνδεσιμότητα, με πλοία ή σειροδρόμους που βρίσκονται εν κινήσει, κάτι που δυσκολεύει τον φύλακα να συμβουλευτεί το σύστημά του. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην, στον αριθμό των θεωρήσεων που εκδίδονται και εκείνων που ελέγχονται στα σύνορα. Το 2015 και 2016 οι πέντε χώρες Σέγγεν που είχαν εκδώσει τον μεγαλύτερο αριθμό θεωρήσεων είχαν ε, κάνει πολύ λιγότερους ελέγχους θεωρήσεων από τον αριθμό τον οποίο είχαν εκδώσει. 80 εκατομμύρια ήταν οι ε, θεωρήσεις που είχαν εκδοθεί και 14, 14 εκατομμύρια ήταν οι θεωρήσεις που είχαν ε, ελεγχθεί. Γι' αυτό και χρειάζεται να ληφθούν από την Κομισιόν διορθωτικά μέτρα. Ένα πληροφορικό σύστημα ε, ε και η ισχύ του εξαρτάται μόνο από τα δεδομένα που περιλαμβάνει. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται, ενώ άλλα που, δεδομένα δεν περιλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται μόνο εν μέρη ή δεν υποβάλλονται και δεν εισάγονται εν Επίσης διαπιστώσαμε ότι τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν μόνο τις ε, μικρής διάρκειας ε, θεωρήσεις Σέγγεν και όχι τις άλλες, τα άλλα είδη θεωρήσεων ε, διαμονής που υπάρχουν ακόμα σε κράτη-μέλη και που επιτρέπουν την πρόσβαση στην περιοχή Σέγγεν. Αυτές οι άδειες εισάγονται μόνο σε εθνικές βάσεις δεδομένων και δεν γίνεται κοινοποίηση της προς άλλους χώρες. 2,6 εκατομμύρια θεωρήσεις ε, εκδόθηκαν το 2016 στην ε, περιοχή Σέγγεν. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την ένταξη αυτών των θεωρήσεων και αυτών των αδειών στο ΒΙΣ. Έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα, γι' αυτό και εμεί δεν έχουμε υποβάλει συγκεκριμένη σύσταση ω προ αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ε, ανάγκη να ε, υπάρξει επικέντρωση στην ποιότητα των δεδομένων που εισάγονται στο πρόβλημα και γι' αυτό καλούμε την ε, Κομισιόν να βελτιώσει τη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων. Ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη βελτίωση των συστημάτων είναι η έγκαιρη υποβολή και εισαγωγή των στοιχείων. Και τα δύο αυτά, και η ποιότητα και ο έγκαιρος χαρακτήρας υποβολής των δεδομένων επηρεάζει την ποιότητα των συστημάτων αυτών. Για παράδειγμα, έχουμε τη διαβίβαση των δακτυλικών ε, αποτυπωμάτων στη Eurodac. Από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Eurodac, δεν, δεν έχει υπάρξει ούτε μία χρονιά κατά την οποία όλα τα κράτη-μέλη να έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ε, έγκαιρα. Το 2015 πάνω από το 50% της, ε, των περιπτώσεων διαβίβασης Eurodac στην, δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Eurodac περέβαιναν το όριο των 72 ωρών που έχει προβλεφθεί. Ε, αυτό ε, το διαπιστώσαμε ιδίως στην Ισπανία. Γι' αυτό και καλούμε την Κομισιόν να ελέγξει αυτές τις ε, ε, περιττές καθυστερήσεις που διαπιστώσαμε και καλούμε την Κομισιόν να λάβει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. κυρία Πέγκοβα είναι η Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γιάκοψεν για την παρουσίαση. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή είναι αρκετά χρήσιμη και ενημερωτική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις συστάσεις που δώσατε, οι οποίες βασίζονται στα πορίσματά σας. Κάποια γενικά σχόλια θα ήθελα να κάνω και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ε, προφανώς. Και ε, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια θα έπρεπε να τεθούν απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι σε εσά. Καταρχά, στην τελευταία σα παρατήρηση αναφερθήκατε στο πώς διατηρούνται τα στοιχεία στο σύστημα πληροφορικής. Ε, ξέρω ότι αυτό ισχύουν ε, ε, για τις χώρες Σέγγεν και τις υποψήφιες χώρες Σέγγεν και ένα από τα βασικά συμπεράσματα τα οποία μας είπατε είναι ότι δεν δίνονται πάντα τα στοιχεία γέρος και δεν χρησιμοποιείται το σύστημα πλήρως όσο θα μπορούσε. Θα ήθελα να, λοιπόν να μου πείτε την άποψή σας και πώς θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να ε, έχει αντίκτυπο στα κράτη-μέλη και στις χώρες που είναι υποψήφιες για να ενταχθούν στο σύστημα Σέγγεν αν δεν λαμβάνουν ε, ε, όλες τις πληροφορίες που διατίθεται στο σύστημα. Παραδείγματο χάρη, έστω ότι υπάρχει μια σημαντική πληροφορία για κάποιον ο οποίος έχει κάνει αίτηση ασύλου. Πώς μπορεί η υποψήφια χώρα Σέγγεν να δράσει καταλήλως. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και θα ήθελα να σχολιάσετε αυτή. Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει και κάποιο αντίκτυπο για τις υποψήφιες χώρες. Και η επόμενη ερώτηση είναι ότι γνωρίζω ότι στην έκθεση αναφέρεστε σε ε, δύο ε, επιπλέον συστήματα πληροφορικής, το σύστημα εισόδου-εξόδου και το σύστημα ταξιδιωτικών πληροφοριών και έγκρισης. Και αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει εντός του 2020-2021 να ξεκινήσει η εφαρμογή τους. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε πληροφορίες ε, επιπλέον για την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ε, φαντάζομαι ότι δεν είναι απαραίτητο ότι έχετε τις πληροφορίες, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αν έχετε όμως κάποια εικόνα για το τι γίνεται, τι χρηματοδοτικοί πόροι χρειάζονται για αυτό το σύστημα κλπ. Και φυσικά υπάρχουν περισσότερε ερωτήσει τι οποίε πρέπει να απευθύνουμε κυρίω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, ε, για την ε, χρηματοοικονομική διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων, δεδομένου ότι τα θέματα προστασία και ελέγχου των συνόρων είναι μία από τι βασικέ προτεραιότητες στο επόμενο ΠΔΠ. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ και πάλι για τα απορίσματα και τι συστάσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Τζετελίνα ε, πρέπει να φύγει. Σας παρακαλώ λοιπόν να τις απαντήσετε, γιατί δυστυχώς ε, το αεροπλάνο δεν θα την περιμένει. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Πένκολα Ναι, φυσικά. αν κατάλαβα καλά, ρωτάτε τι γίνεται αν δεν συμπεριληφθούν τα δεδομένα στα, ε, στο σύστημα και τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Αναφέρεστε σε υποψήφιες χώρες, η Κομισιόν πρέπει να απαντήσει γι' αυτό, αλλά για τα κράτη-μέλη της Σέγγεν ε, πρέπει να πω ότι, όπως δείχνει και η έκθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαθέτουμε τις πληροφορίες, να τις ανταλλάσσουμε και να τις χρησιμοποιούμε για την προστασία των εξωτερικών συνόρων όταν δεν τροφοδοτούνται τα συστήματα με τα απαραίτητα ε, στοιχεία ε, και σε επίπεδο ποιότητας αλλά και γέρος τότε αυτοί οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια τελικά μπαίνουν στο σύστημα Σέγγεν χωρίς ε, να γίνει το κατάλληλο έλεγχο. Και επομένω υπάρχει κίνδυνο τρομοκρατία, εγκλήματο, αλλά και η απέτηση κάθε χώρα Σέγγεν να γνωρίζει ποια άτομα βρίσκονται στην επικράτειά τη. Εάν δεν διαθέτει κάποιο τα στοιχεία για να κάνει συγκριτική ανάλυση, σημαίνει ότι δυσχεραίνεται και το έργο των συνοριοφυλάκων όσον αφορά τα νέα συστήματα, σωστά θα εφαρμοστούν νέα συστήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το που βρισκόμαστε και όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται. Όπως βλέπετε και από τη δική μας την έκθεση, εμείς λέμε ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, αλλά ήταν ε, αργή απορρόφηση γιατί είναι επαχθής η διαδικασία λόγω των διαφόρων κανονισμών, θέματα ανταγωνισμού, ε, για να ξεκινήσει κάποιο να αντλεί τους οικονομικούς πόρους. Ε, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να απευθύνετε απευθεία ε, το ερώτημα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης του ΕΛΚ. Μέρς. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω πτήσει να πάρω. Ευχαριστώ το συνέδριο για τη στήριξή του. Η έκθεση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και είναι και επίκαιρη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναπτύξουμε την διαλειτουργικότητα των διαφόρων στοιχείων του συστήματος. Άρα καλό είναι να δούμε και πόσο αποτελεσματικά είναι. Χαίρομαι που οι συνοριοφύλακες τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο και ότι είναι καλά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τους συνοριακούς ελέγχους. Αλλά εκφράζω και μια σειρά ανησυχίες, να αναφερθώ σε ορισμένες, δακτυλικά αποτυπώματα. Και η δυνατότητα βιομετρικών ελέγχων. Μόνο 10 κράτη Σέγγεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Άρα είναι πιο πολύ ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ είναι δυνατόν να είναι έτσι η κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπιστεί. Διότι αυτό οδηγεί και σε κάτι άλλο που εντοπίζει η έκθεση, ότι οι συνοριοφύλακε ορισμένες φορές έχουν πολλά ε, ε, ε, λανθασμένα θετικά και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι η χρήση ε, του βιομετρικού ελέγχου. Επίσης η ερμηνεία του κανονισμού ΣΥΣ. Πώς γίνεται. Η Γαλλία δεν τα χρησιμοποιεί για να ε, ζητάει καταλόγους επιβατών. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν μια χώρα δεν χρησιμοποιεί τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων για να ελέγχει τους επιβάτες, αυτό θα ήταν μια δυναμία σε όλο το περιβάλλον ασφαλείας μας. Είπατε ότι δεν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη γιατί είναι βαριές οι διαδικασίες προμηθειών και καθυστερούν. Τι μπορούμε να αλλάξουμε. Θεωρείτε ότι είναι υπερβολικά βαριές οι διαδικασίες, δηλαδή ότι ακατάλληλες για το στόχο τους. Έχουμε τα χρήματα και δεν τα αξιοποιούμε. Είναι κρίμα, ιδιαίτερα για το ISF. Αυτό που με ανησύχησε περισσότερο είναι ότι μισοί συνοριοφύλακες είπαν ότι χρειάστηκε να επιτρέψουν σε κάποιον ε, να μπει στο χώρο Σέγγεν χωρί να ελέγχουν τα στοιχεία του. Και είπατε ότι αυτό γίνεται, ορισμένοι συνοριοφύλακε είπαν ότι γίνεται συχνά. Θεωρείτε ότι είναι επαρκώ αντιπροσωπευτικό το δείγμα για όλη την Ένωση. Και μα ανησυχεί αυτό το θέμα. Ω Κοινοβούλιο είχαμε ένα ψήφισμα και έκθεση πέρυσι για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν Άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και πάλι στρέφουμε προς την Κομισιόν. Για το μηχανισμό αξιολόγησης λειτουργίας του Σέγγεν. Στο ίδιο ψήφισμα συμφωνούμε πολύ ότι οι επιπτώσεις, τα μέτρα που λαμβάνονται μετά τις αξιολογήσεις, λαμβάνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τι πρέπει να αλλάξει για να γίνονται οι αλλαγές αλλά και το σύστημα αυτών των ε, αξιολογήσεων. Ε, αναφερθήκατε μόνο στις ε, προαναγγελθήσεις επισκέψεις. Η έκθεση της Κομισιόν μιλάει και στις, για τις εξαπίνεις. Και αυτές ακόμη οι εξαπίνεις σε ένα βαθμό δεν είναι τόσο εξαπίνεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας το εξηγήσει. Ακόμη και αν πάτε χωρίς να το έχετε πει, το κράτος μέλος μαθαίνει ότι θα γίνει μια αξιολόγηση. Είναι όταν ήμουν φοιτητή, α πούμε, όταν μου είχε πει η μαμά μου ότι θα έρθει, συγύριζα το δωμάτιό μου. Ε, έτσι κάνουν και τα κράτη-μέλη. Τώρα είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, δεσμευτικές προθεσμίες για το Eurodac. Κοιτάξτε, όταν τα συζητάμε, το Κοινοβούλιο θέλει πιο αυστηρές προθεσμίες και το Συμβούλιο λέει «Μα δεν είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο». Και καταλήγουμε σε διατυπώσεις του τύπου όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς καθυστέρηση. Βοηθάνε τέτοιες διατυπώσεις για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Στο νέο αναθεωρημένο κανονισμό ΣΥΣ λέει σε διάφορα σημεία χωρίς καθυστέρηση, χωρίς καθυστέρηση και στην πράξη αυτό σημαίνει καθυστέρηση. Για την ποιότητα των στοιχείων αναφερθήκατε στο ΣΥΣ. Κοιτάξτε, ορισμένες φορές ε, σε ποινικέ περιπτώσεις. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία που θα θέλαμε, αλλά βάζουμε ό,τι έχουμε, γιατί είναι καλύτερα από το τίποτα. Στα, στις άλλες βάσεις ε, στοιχείων ε, πώς αξιολογείτε την ποιότητα των στοιχείων. Η αξιολόγηση είναι πολιετής. Είδατε τον αναθεωρημένο κανονισμό για το ΣΥΣ και τον κανονισμό για την διαλειτουργικότητα. Γιατί ανησυχείτε στην έκθεσή σας ότι το EU Λίζα και η Επιτροπή δεν έχουν επαρκείς κανόνες για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων. Νομίζω ότι αυτά τα δύο που προανέφερα βελτιώνουν το ρόλο του Λίζα και της Επιτροπής. Έχετε σχόλια. Και βεβαίως το Συμβούλιο δεν είναι παρόν, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι ακούγεται περίεργα το ότι το Συμβούλιο για το επόμενο πλαίσιο θέλει να δώσει 7,5 δις λιγότερα από τις προτάσεις της Κομισιόν για τους ελέγχους των συνόρων και τη μετανάστευση. Αν θέλουμε να έχουμε σωστούς ελέγχους ε, των συνόρων, πρέπει να ε, δαπανίσουμε και τα ε, απαραίτητα ποσά. Ευχαριστώ, Ολιβιέ Σαστέλ. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω το συνέδριο. Μια εκθεσία αυτή είναι σημαντική, ενδιαφέρουσα. Η παρουσίαση ήταν πολύ ενημερωτική. Πρώτα απ' όλα πώς ε, λειτουργούν και πώς άλλοι λεπιδρούν τα διάφορα συστήματα πληροφόρησης για να βοηθήσουν τους συνοριοφύλακες. Και συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες του συνεδρίου Πώς δηλαδή μπορούν να μπουν οι συνοριοφύλακες ε, στο σύστημα δεύτερης γενιάς, ότι δεν περιέχει όλα τα στοιχεία και ότι δεν το γνωρίζουν και αρκετά καλά αυτό το σύστημα. Γενικά οι περισσότεροι. Μας είπαν ότι δεν έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση. Στο χώρο Σέγγεν η πολιτική θεωρήσεων είναι προφανώς κοινή. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι θεωρήσεις που χορηγούνται χορηγήθηκαν σωστά και ότι ο έλεγχος έγινε σωστά με τήρηση όλων των κανόνων. Και λυπούμε που δεν υπάρχει περισσότερη εναρμόνιση των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη για το Eurosur. Μόνο οι μισές ε, ευρωπαϊκές χώρες ανταλλάσσουν πληροφορίες. Ελπίζω οι συστάσεις του συνεδρίου να ε, γίνουν πράξη τάχιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς, κάτι πολύ σύντομο. Έχω την εντύπωση ότι γίνονται πολλά, αλλά ότι το σύστημα έχει ε, τόσες τρύπες όσο η γραβιέρα Ελβετίας. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό δεν μπαίνω σε επιμέρους τώρα ερωτήσεις. Είναι πολύ ζώρικη η κατάσταση. Ωραία. Θέλει κανείς άλλος τίποτα. Όχι, ωραία. Να δώσω το λόγο στο συνέδριο. Ευχαριστώ. Απλώς να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που τέθηκαν και από εκεί και πέρα θα, δώσω, θα αφήσω ε, την Κομισιόν να απαντήσει. Πράγματι, υπάρχουν διάφορες νομικές ερμηνείες για τους κανόνες που πρέπει κανείς να τηρήσει Κάτι που μπορεί να δημιουργεί μια μικρή έκπληξη, αλλά αυτό προέκυψε από τον έλεγχο που κάναμε. Μας ε, ε, ρωτήθηκα για τους ε, επαχθείς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Πάντοτε είναι ωραίο σύνθημα η απλοποίηση, αλλά είναι ζητούμενο και δύσκολο εγχείρημα το να απλοποιήσει κανείς τους, τους κανόνες. Πολλές συχνά τα κράτη-μέλη δηλώνουν ότι είναι δύσκολη η, κανο... η τήρηση των κανόνων. Φυσικά δεν είναι μόνο... οι συνοριοφύλακε, δεν χρησιμοποιούν μόνο τα πληροφορικά συστήματα, χρησιμοποιούν την εμπειρία του, την τεκμηρίωση που έχουν στη διάθεσή του, τα έγγραφα προφανώ που υποβάλλονται, ε, έχουν λάβει εκπαίδευση ε, όσον αφορά τα παραποιημένα έγγραφα. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα θα πρέπει να εισάγονται έγκαιρα και με πλήρη τρόπο ώστε να υποστηρίζουν τους συνοροφύλακες στη δουλειά τους από, την, από το δείγμα μας τα 951 άτομα που ρωτήσαμε ε, νομίζω ότι το δείγμα αυτό είναι αντιπροσωπευτικό ε, προ, προέρχονταν οι και από όλα τα κράτη-μέλη οπότε νομίζω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό το δείγμα. Σχετικά με τις καθυστερήσεις θα έλεγα ως ελεγκτής ότι είναι πάντοτε καλύτερο να υπάρχει μια συγκεκριμένη προθεσμία, μια συγκεκριμένη ημερομηνία να λέει δηλαδή κανείς ότι ε, μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Πάντοτε καλύτερο από το να λες σύντομα ή εν ευθέτω χρόνο κτλ. κτλ. Οπότε είναι μια σύσταση προς την Κομισιόν να το λάβει σοβαρά υπόψη τη. Ε, ελβετικό τυρί. Διάτριτο σύστημα είπατε. Όταν έχει κανείς πληροφορικά συστήματα που πρέπει να συνεργαστούν. Υπάρχουν πάντοτε προβλήματα διαλειτουργικότητας, συνδεσιμότητα, αν θέλετε. Βεβαίως στην πορεία είμαι βέβαιη ότι η Κομισιόν θα προσπαθήσει να βελτιώσει ε, τα συστήματα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να συγχωνεύουμε όλα τα δεδομένα και να υπάρχει μια καλή ροή των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων. Σχετικά με το πώς εξασφαλίζουμε ότι οι θεωρήσεις εκδίδονται με ενιαίο και ομοιογενή, ε, τρόπο. Υπάρχουν ακόμα 100 δυνατότητε εθνικές για την έκδοση θεωρήσεων, όπως το παράδειγμα που σας έδωσα στην, ε, στην παρουσίασή μου. 2,6 εκατομμύρια ε, διαφορετικές θεωρήσεις εκδίδονται στην περιοχή στην περιοχή Σέγγεν που δεν μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών. Και η αναγνώριση, η Κομισιόν μάλλον έχει αναγνωρίσει ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι θεωρίες δεν μπορούν να ε, ε, εισάγονται στο ΣΥΣ. Έχει αναγνωρίσει αυτό το πρόβλημα και ε, νομίζω ότι και από τη σκοπιά ενός ελεγκτή είναι εμφανές και προφανές το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μαζί μας την ε, Μάγδα Τσίγκαν από την ε, Κομισιόν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει την εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, την κυρία Γιάκοψεν και την ομάδα ελέγχου της για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στη διαδικασία αυτή ε, στη διάρκεια των μηνών που χρειάστηκαν προκειμένου να εκπονηθεί η έκθεση. Χαιρόμαστε για την έκθεση που υποβλήθηκε σήμερα στην Επιτροπή σας, διότι αποτελεί και αναγνώριση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθούν και να υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη για να κάνουν πιο αποτελεσματικούς ελέγχους στα σύνορα, χρησιμοποιώντας ε, τα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρόμαστε επίσης που μας δίνετε και την ευκαιρία για αλλαγή απόψεων και έχω ήδη συλλέξει αρκετά σχόλια και ερωτήσεις ε, για τη συζήτηση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το συνέδριο έκανε κάποιες ε, θετικές παρατηρήσεις που είναι πολύ σημαντικές για μας ε, και σας ευχαριστούμε και καταρχάς ότι είναι καλός ο σχεδιασμός των συστημάτων για να διευκολύνουν τους έλεγχους στα σύνορα και στα κράτη-μέλη σε γενικές γραμμές συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει επίση αναγνώριση του μηχανισμού εξιολόγησης Σέγγεν ω μηχανισμό, ω μια δομή που ε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και φυσικά υπάρχουν θέματα μεθοδολογίας και βασικών τυχών του συστήματος. Τα κράτη-μέλη που είναι πολύ σημαντικός παράγον στην όλη διαδικασία και στα όλα θέματα εφαρμογής χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ε, τα βασικά συστήματα πληροφορικής και βασίζονται σε αυτά ε, κατά την εκτέλεση των ελέγχων στα σύνορα και ε, μοιράζονται όλο και περισσότερες πληροφορίες μέσω των συστημάτων. Η έλεγχη στα σύνορα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, καλύπτουν μεγάλο σκέλος των πολιτικών μας και θα ήθελα επίσης να επιστήσω και την προσοχή σας στο γεγονό ότι το ελεγκτικό συνέδριο έκανε μία πληρέστατη έρευνα και ανάλυση, διότι το θέμα αφορά και τα ε, συστήματα πληροφορικής ε, αυτά καθεαυτά, το SIS και το VIS, αλλά και το EuroShare και το PNR που εξηγούνται πάρα πολύ καλά, δίνεται και περιγραφή των συστημάτων στην έκθεση. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά, γιατί αναφέρονται και στην πρακτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Εδώ ε, αναφέρομαι στο Eurosur, που δεν είναι μόνο ένα σύστημα πληροφοριών το οποίο είναι συγκρίσιμο με το SIS και το VIS, αλλά είναι και μία πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και του Frontex. Και όσον αφορά το PNR, το σύστημα των στοιχείων των επιβατών, η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αυτή η οποία δεν δημιουργεί ένα κεντρικό σύστημα πληροφορική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα συλλέγονται βάσει τη οδηγία PNR όμω και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπού επιβολή του νόμου. Είναι πολύ σημαντικά και αυτά τα στοιχεία και χρειάζονται για να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση. Όπως σας είπα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις θετικές ε, αξιολογήσεις, αλλά φυσικά ε, χαιρόμαστε και ιδιαίτερα με τις συστάσεις. Όλες αυτές οι συστάσεις είναι αποδεκτές από μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τις εφαρμόσουμε εντός των πλαισίων της εντολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε την εφαρμογή των συστάσεων μεταξύ των κρατών μελών και των οργανισμών και υπηρεσιών που ε, μπορεί να ε, τις αφορά. Να απαντήσω τώρα και σε κάποια από τα σχόλια. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις, διότι πρέπει ε, να σχολιάσουμε όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα σαφές πλαίσιο για τη χρήση των συστημάτων. Ε, τα κράτη-μέλη, οι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα η Αστυνομική Ακαδημία, ε, η ΣΕΠΟΛ, ε, που είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των αστυνομικών, και το EU LISA, που είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια, έχουν κάνει τη σημαντική ανάλυση σε θέματα κατάρτισης και ασφάλειας. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Γιουλίζα θα αξιολογήσει βάσει των συστάσεων και των παρατηρήσεων του δικαστηρίου τη χρήση τη βασική κατάρτιση καταρχά ε, από πλευρά κρατών μελών και θα συνεχίσουμε να του προτρέπουμε να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε ήδη. Τα κράτη-μέλη παρεμπιπτόντω εξετάζουν όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο ε, την επένδυση σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ε, ε κατάρτισης στο διαδίκτυο και επίσης υπάρχει και η νομοθεσία η οποία καθορίζει τα σχετικά συστήματα πληροφορικής που θα δώσει τη δυνατότητα στο Frontex να αναπτύξει συγκεκριμένες διαπαφέ, οι οποίες θα είναι χρήσει ε, κατάλληλες ε, για τους ε, αξιωματικούς που θα είναι ε, φιλοξενούμενοι σε σημεία συνόρων σε άλλε χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα επηρεάσει και το έργο μα με το ελεγκτικό συνέδριο επί της ε, πτυχή αυτή. Όσον αφορά τι ελλείψει που διαπιστώθηκαν κατά τις αξιολογίες τη έννοια, επειδή δεν υπάρχουν δεσμευτικέ προθεσμίε. Ε, συμφωνούμε κατ' ουσίαν με την ε, άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου και εδώ χρειαζόμαστε πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αλλά εμείς από πλευράς μας εξετάζουμε και διαδικαστικές και πρακτικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν συνολικά το χρόνο ε, κύκλου αξιολόγησης Σέγγεν. Το επόμενο σημαντικό βήμα επ' αυτού είναι ότι ο κανονισμός Σέγγεν προβλέπει υποχρέωση αναθεώρησης του μηχανισμού μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου και η αξιολόγηση αυτή θα γίνει το 2020. Επομένως θα είναι και μια καλή ευκαιρία να δούμε ε, τη σύσταση αυτή στο πλαίσιο αυτό καθυστερήσεις για την εφαρμογή λύσεων πληροφορικής, ιδέως ε, για το Eurosur και το PNR σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πράγματι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις ε, για τις ε, λύσεις πληροφορικής για το Eurosur, αλλά δεν ήταν και πολύ μακρές οι καθυστερήσει. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Είναι απλώ μια περιγραφή της κατάσταση στην πράξη. Όπως είπα και στην αρχή, το Eurosure δεν είναι μόνο ένα σύστημα δεδομένων, είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας. Και αυτό το δίκτυο επικοινωνίας διασυνδέει τα κράτη-μέλη, τα δίκτυα και τα κέντρα συντονισμού για την εποπτεία των συνόρων και το Frontex και επομένως έγινε γέρος και επιτρέπει για παράδειγμα την ανταλλαγή πληροφοριών για ε, περιστατικά που αφορούν παράτυπη μετανάστευση και διασυνοριακό έγκλημα. Αλλά πράγματι υπήρξε καθυστέρηση στη δημιουργία του συνολικού συστήματος και μάλιστα ήταν και μια ε, σύνθετη διαδικασία ε, πιστοποίησης στα κράτη-μέλη για την ανταλλαγή κάποιων πληροφοριών λόγω θεμάτων εμπιστευτικότητας. Υποστηρίζουμε φυσικά και τα κράτη-μέλη για να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, αλλά πράγματι είναι ένα από τα στοιχεία αυτά η πλήρης διαδικασία πιστοποίησης και η πλήρη ως έλεγχος ασφαλείας των ατόμων που συμμετέχουν σε θέματα εμπιστευτικότητας, που ε, είναι αμυγός ε, στα χέρια των κρατών μελών. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή για το PNR, αυτή τη στιγμή 26 κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει ότι έχουν μεταφέρει τους κανόνες του PNR στην εθνική τους νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζει ενεργά τα κράτη-μέλη στη διαδικασία εφαρμογής ε, παρέχοντας ε, τη χρηματοοικονομική στήριξη για την αγορά του απαραίτητου hardware και λογισμικού καθώς επίσης και βοηθά με συντονισμό, με τακτικές συνεδριάσεις ε, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και φυσικά θα το συνεχίσουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτή τη στήριξη και την καθοδήγηση ώστε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως ε, και σωστά τους κανόνες. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι και σχετικά πρόσφατο εργαλείο της προηγούμενης χρονιάς και αυτό είναι αντικειμενικό, αλλά έπρεπε να λάβουμε υπόψη και κάποια στοιχεία όταν ε, γινόταν η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και κυρίως το γεγονός ότι το να υπάρχει συνδεσιμότητα με τις αεροπορικές γραμμές είναι αρκετά περίπλοκο και ορισμένες φορές σε κάποιες περιπτώσεις ε, χρειάστηκαν και 6 έως 9 μήνες για την κάθε αεροπορική εταιρεία. Η διαδικασία βέβαια είναι σε εξέλιξη, προχωράει και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν την οδηγία. Κάτι πολύ ενδιαφέρον για τα κενά στους ελέγχους ε, των θεωρήσεων στα σύνορα και των θεωρήσεων που εκδίδονται. Εδώ λαμβάνουμε υπόψη τη σύσταση και θα δούμε γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα αναλυτικά σε σχέση με τον αριθμό των θεωρήσεων που εκδίδονται και αυτών που ελέγχονται στα σύνορα και αν χρειαστεί θα προτείνουμε διορθωτικά μέτρα. Ε, ίσως ε, έχει σημασία και θα έπρεπε να υπενθυμίσω και λίγο το πλαίσιο αυτών των ελέγχων μεταξύ του 2015 και του 2017 είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος αναφοράς. Πέντε χώρες αναφέρονται εδώ και ε, όπως και να έχει όμως ε, θα το εξετάσουμε πιο εκτεταμένα. Τώρα, για την ποιότητα των δεδομένων, εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα του SIS και δεν μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση κάθε ε, περίπτωσης ξεχωριστά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό που εξασφαλίζουμε είναι ότι υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί και δικλείδες ασφαλείας στα κράτη-μέλη ή για να έχουμε υψηλής ποιότητας δεδομένα στο σύστημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γιουλίζα είναι στη διαδικασία βελτίωσης αυτών των μηχανισμών για την παρακολούθηση την ποιότητα των δεδομένων και το θέμα αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τακτικά και συζητάται στη σχετική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, η Επιτροπή SIS-VIS και υπάρχουν και κάποια εργαστήρια για την ποιότητα των δεδομένων που διοργανώνονται για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτά ε, για τις συστάσεις και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλή στιγμή για να έχουμε αυτές τις στάσεις, είναι κατάλληλα στοχευμένες, βασίζονται στην αξιολόγηση της κατάστασης και εμείς ε, στα πλαίσια της εντολής μας και με τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς θα συνεργαστούμε προκειμένου να τις εφαρμόσουμε. Ε, ένα-δυο στοιχεία ακόμα από τη συζήτηση να φίξω για τις ευνηδιαστικές επισκέψεις. Πράγματι, το σχολιάσαμε αυτό στην έκθεση του ελεγκτικού ε, δικαστηρίου, πέραν από τους τακτικούς ελέγχους, υπάρχουν και αρκετές ε, ε, ευνηδιαστικές επισκέψεις στη διάρκεια του έτους και σε αυτές τις επισκέψεις μπορούμε να εξετάσουμε κατά πόσο εφαρμόζονται προηγούμενες συστάσεις και Έχουν υπάρξει ευνηδιαστικές επισκέψεις και αρκετές ε, επαναληπτικές επισκέψεις όταν γίνεται για να εφαρμοστεί κατά πόσον ε, να εξεταστεί κατά πόσον συγγνώμη εφαρμόστηκαν οι προηγούμενες συστάσεις. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία και των ε, ε τακτικών ελέγχων αλλά και των ευνηδιαστικών επισκέψεων είναι για να μπορέσουμε να ελέγχουμε τη διαδικασία και να έχουμε κατά νου και το τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό θα συζητηθεί βεβαίως πιο διεξοδικά από τους ε, αρμοδίους ε, στο μέλλον. Να επιστήσω και την προσοχή σας στο γεγονό ότι εντός της εβδομάδας αυτής ε, τέθηκαν σε ισχύ αλλαγές για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή και πλέον θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή αυτών των νέων λύσεων και κυρίως ε, τη δέσμη μέτρων για τη διαλειτουργικότητα, αλλά και το EPCG που περιλαμβάνει μια σειρά από στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά πλέον με την έναρξη ισχύω και νομίζω ότι για τα μελλοντικά ε, στοιχεία την εφαρμογή του Entry Exit, του συστήματος εισόδου-εξόδου και του ETIAS. Ε, ε, μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση για κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν. Επομένως θα μπορέσουμε να δούμε ε, θεωρητικά κάποια πράγματα, αλλά θα λάβουμε υπόψη και τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό το ελβετικό τυρί και να γίνει παρμεζάνα. Κάτι τέλος πάντων χωρίς τρύπες. και να μην έχει τα κενά τα οποία διαπιστώσαμε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Grazie, grazie. Σας ευχαριστώ πολύ για τις περαιτέρω διευκρινήσεις, οι οποίες ήταν πληρέστατες. Η κυρία Γιάκοψεν από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ήθελε να προσθέσει κάτι ακόμα μετά από αυτά που ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείτε ότι έχετε κάτι να προσθέσετε. Αν ναι, ναι, να σας δώσω το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Όπως είπα, ένα σύστημα πληροφορικής ε, είναι τόσο καλό όσο τα στοιχεία που περιέχει. Σημαντικό είναι λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τα συστήματα αλλά και ότι η φύση και το είδος των στοιχείων που περιέχουν βελτιώνονται. Είναι καλό το σύστημα αυτό. Βοηθάει πολύ τους νεροφυλακές που κάνουν ε, καλά τη δουλειά τους, αλλά χρειάζονται και καλά συστήματα προφορικής. Εξαρτώνται όλο και περισσότερο από αυτά. Πρέπει να εστιάσουμε στην έγκαιρη εισαγωγή πλήρων στοιχείων. Και αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία θέλω να το επιβεβαιώσω και εγώ. Ήταν θαυμάσια συνεργασία μας κατά τον έλεγχο. Θέλω τον, ε, να τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική τους, να τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική τους συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς κυρία Γιάκοψεν. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο και τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Την ειδική έκθεση 24 του 2019 για το άσυλο και τη μεταγκατάσταση και την επιστροφή μεταναστών. Να δώσω αμέσως ε, το λόγο στον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Μπρινκάτ, τον οποίο και καλωσορίζω. Σας δίνω το λόγο για την παρουσίαση για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Thank you, Madam, Madam Chair. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα για την ε, ευγενική σας πρόκληση. Θα σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για το θέμα αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε το χάσμα μεταξύ στόχων και αποτελεσμάτων. Μαζί με, τα ε, με τις ε, απαντήσεις της Κομισιόν και όσα μας είπε η Φράντεξ και η Άσο. Τα τελευταία χρόνια στην Ένωση έχουμε πρωτόγνωρα ποσοστά ε, αιτήσεων ε, μετανάστευσης και ασύλου. Το 2017 δημοσίευσαμε την έκθεση για τα hot spot που, hot που δημιουργήθηκαν στην ε, Ιταλία και την Ελλάδα για να είναι ο πρώτος χώρος υποδοχής όπου ταυτοποιούνται, καταγράφονται και λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτελέσματα των μεταναστών. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα πόρισματά μας αλλά μας ζήτησε να κάνουμε και μία ανάλυση του συστήματος μετεκατάστασης, ασύλου και επιστροφών. Η έκθεση λοιπόν αυτή θα έλεγα είναι μια υβριδική έκθεση. Είναι και ε, συνέχεια του συστηματος μετεκατάσταση ασυλου και επιστροφων η εκθεση λοιπον αυτη θα ελεγα ειναι μια υβριδικη εκθεση ειναι και συνεχεια του ενεχου μα στα hotspot και αφορά την μετανάστευση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και τη διαχείρισή της. Κυρίως εξετάζουμε εάν ε, επιτύχαμε τους στόχου που επιδιώκαμε χρηματοδοτώντα την Ιταλία και την ε, Ελλάδα και αν ήταν ε, αποτελεσματικέ και ταχείε οι παρεμβάσει μα. Και επίση εξετάσαμε ε, και κατά πόσο τα προσωρινά συστήματα μετεκατάσταση επέτυχαν του στόχου του. Όπω ξέρετε πολύ καλά, το ελεκτικό συνέδριο δεν διαμορφώνει πολιτική. Οι έλεγχοί μα έχουν να κάνουν με τη χρηστή χρήση των πόρων. Γιατί είμαστε θεματοφύλακε των οικονομικών. Και τονίζω ότι η εργασία μας ολοκληρώθηκε πριν το περασμένο καλοκαίρι. Ένα άλλο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι στι αρχέ του 2019, όταν οι τεχνικέ μα ομάδε έκαναν τον έλεγχο, άκουσα τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και όσων ασχολούνται με το θέμα αυτό. Είχα συναντήσεις με πολλούς ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο και αυτό μου επέτρεψε να καταλάβω καλύτερα το θέμα. Κάτι που θα κάνω και για τον έλεγχο που κάνουμε τώρα της ε, Frontex, ε, του οποίου ηγούμε. Τώρα για την ειδική έκθεση. Καταλήγουμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους στόχους της ε, Ένωσης και τα αποτελέσματα που επιτυχάνονται. Παρά το ότι οι δυνατότητες στην Ιταλία και την Ελλάδα βελτιώθηκαν, η εφαρμογή των διαδικασιών ασύλου στην Ιταλία και την Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στενώσεις οι επιστροφές από την Ελλάδα και την Ιταλία είναι χαμηλές. Όπως λέμε και στα απορίσματά μας θεωρούμε ότι οι συστάσεις μας ε, της ειδική έκθεσης του 2007 είχαν εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό ή ήταν ε, σε φάση εφαρμογής και είπαμε που αυτό δεν γίνεται. Παρά το ότι η καταγραφή και η λήψη αποτυπωμάτων έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα στα hotspot, παρόλα αυτά τα προσωρινά ε, προγράμματα Μετεκατάσταση δεν επιτυχάνουν του στόχου, άρα δεν μειώνεται η πίεση στο σύστημα στην Ιταλία και την Ελλάδα. Εξετάσαμε 20 δράσει στήριξη τη Ένωση στην Ελλάδα και την Ιταλία και παρά το ότι εντοπίζουν τις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει, υπάρχουν αδυναμίες στο σχεδιασμό του. Επίση διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα προγράμματα που εξετάσαμε δεν είχαν επιτύχει πλήρω τους στόχου του. Ε, αξιολογήσαμε το πλαίσιο διαχείρισης και θεωρήσαμε ότι δημιουργήθηκε αργά και χωρίς στόχους. Κάτι πιο ανησυχητικό, δεν είχαμε επαρκή στοιχεία για τις επιδόσεις των προγραμμάτων. Αξιολογήσαμε την επίπτωση των ε, δράσεων στήριξης της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο εξετάζοντας εάν οι διαδικασίες ασύλου και επιστροφών έχουν γίνει ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές. Διαπιστώσαμε ότι η δυνατότητα ε, εξέτασης περιπτώσεων ασύλου αυξήθηκε και στην Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά όχι επαρκώ για να αντιμετωπίσει τι ε, αυξανόμενε καθυστερήσει στην Ελλάδα. Επειδή υπάρχουν λιγότερε νέε αιτήσει στην Ιταλία, οι καθυστερήσει ε, βεβαίω μειώνονται, αλλά υπάρχει ανεπαρκές δυναμικό για να εξεταστούν οι πολλές ε, εφέσεις κατά τη πρώτη απόφαση. Πολύ λιγότεροι μετανάστες επιστρέφουν από τις αποφάσεις επιστροφής που λαμβάνονται, όπως και στην Ένωση γενικότερα. Εντοπίσαμε τους λόγους γι' αυτό. Κυρίως, παίρνει πολύ χρόνο για να εξεταστεί μια αίτηση ασύλου. Δεν υπάρχει επαρκές δυναμικό στα κέντρα κράτησης. Είναι δύσκολη η συνεργασία με τις ε, χώρες προέλευσης των μεταναστών. Ή οι μετανάστες απλώς δραπετεύουν όταν ληφθεί η χώρα, η απόφαση συγγνώμη, να επιστραφούν. Κυρίως ε, ελέγξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΣΟ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Frontex. Επιπλέον, επισκεφθήκαμε εθνικές αρχές, διεθνές και, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εφαρμόζουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση. Πρέπει να πω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία από όλους τους οργανισμούς που ελέγξαμε. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου μας, συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ανεξάρτητους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τα διδάγματα και την εμπειρία για ενδεχόμενο, έναν ενδεχόμενο μηχανισμό εθελούσιας μετεκατάσταση Να ενισχύσουν τη διαχείριση της επίγουσας βοήθειας και των εθνικών προγραμμάτων που υπάγονται στο Ταμείο για το Άσλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη. Να ενισχύσουν τη συνεργασία της ΕΑΣΟ, την συμμετοχή μάλλον του ΕΑΣΟ στις διαδικασίες ασύλου. Να προσαρμοστεί η στήριξη που δίνεται στην Φράντεξ για τις επιστροφές και η χρήση ειδημόνων στα hotspot. Να ενισχυθεί η διαχείριση των εθνικών συστημάτων ελέγχου και να στηριχθούν περαιτέρω οι εθνικές διαδικασίες επιστροφών. Τονίζω ότι η Επιτροπή και οι φορείς αποδέχθησαν πλήρως όλες τις συστάσεις μας. Κατά λίγο, σας ευχαριστώ και πάλι για την ε, ευγενική σας πρόσκληση και με κάθε χαρά να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βρυνκάτη για την παρουσίασή σας. Για ένα θέμα το οποίο πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο και είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία μας είπατε, αλλά μας καθησυχάζει το γεγονός ότι υπάρχει καλή συνεργασία από πλευράς όλων των ε, εμπλεκομένων. Να δώσω τώρα το λόγο για 10 λεπτά επίσης στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνατε και για την προφορική παρουσίαση της ε, έκθεσης εδώ. Συμφωνώ και εγώ με την ε, Αντιπρόεδρο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και σύνθετο πρόβλημα. Αλλά ακριβώ σε αυτά τα περίπλοκα και σύνθετα και ευαίσθητα προβλήματα χρειαζόμαστε ενιαίες απαντήσεις. Η ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου καταδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η πολιτική μετανάστασης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί κανείς να γνωρίσει ως ε, πολιτική φιλική προς το άσυλο και τους ετούντες άσυλο δεν απέφερε τους επιθυμητούς καρπούς. Όταν προσδιορίσαμε και θεσπίσαμε αυτή την πολιτική ε, ήταν ήδη σαφές ότι κινούμασταν ε, σε λάθος κατεύθυνση και στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην Ολομέλεια έχουν γίνει πάμπολες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Οι συμβολικές αυτές συζητήσεις στις συζητήσεις αυτές κέρδισαν εκείνοι που είναι υπέρ της ε, μετανάστευσης και του ασύλου και ότι θα πρέπει να, καταπολεμήσει, να καταπολεμηθεί η παράτυπη, η παράνομη μετανάστευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όταν τα κράτη-μέλη λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των ε, συνόρων, τότε αυτό οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα και ότι σημαντικότατος στόχος ήταν το κλείσιμο των παράνομων οδών και διαδρόμων εισόδου παράτυπων μεταναστών. Δεν ήταν η κουλτούρα ε, της φιλοξενίας που οδήγησε στην εξομάλυνση της κατάστασης, ήταν το κλείσιμο των παράνομων διαδρόμων μετανάστευσης στα Βαλκάνια και στη Μεσόγεια. Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία έτσι όπως έχουν καταγραφεί στην ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Στην Ιταλία, βάσει των ε, ισχυών των κανόνων, όταν κανείς υποβάλλει αίτηση ασύλου, λαμβάνει υποχρεωτικά απάντηση εντός 33 ημερών. η περίοδος αυτή το 2015 επεκτάθηκε στις 264 64 μέρες, ενώ το 2018 ε, ανήλθε σε πάνω από 400 μέρες χρόνο αναμονής για να τεθεί μια αίτηση ασύλου σε επεξεργασία. Όταν κάποιος παράτυπος μετανάστης λοιπόν εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβάλλει αίτηση ασύλου, αυτό σημαίνει ότι μπορεί η επεξεργασία αυτής της ε, αίτηση να διαρκέσει ακόμα και 437 ημέρες. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα έχει το δικαίωμα να παραμένει στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 437 ημέρες νόμιμα. Αν δεν ε, ε, συνυπολογίσει κανείς και τη διαδικασία εφέσεων, τότε μπορεί να περάσουν ακόμη και ε, χρόνια έως ότου επεξεργαστεί μια αρχή, μια αίτηση τελεσίδικα. Σε ε, πολλές περιπτώσεις, μάλιστα στην Ιταλία, ε, δεν μπορεί κανείς να κάνει λόγο ούτε καν για εκτελεστή απόφαση από τα, από τα δικαστήρια. Όσον αφορά την μετεγκατάσταση, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι Μεγάλο μέρος των ε, ε, ετούντων άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα μπορούν να μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι υποχρεωτική η εισαγωγή των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων στο Eurodac. Από τα στοιχεία λοιπόν που περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι οι μετανάστες ταξιδεύουν με τέτοιον τρόπο ώστε να μην καταγράφονται, να μην λαμβάνονται, να μην καταγράφονται και να μην εισάγονται στο Eurodac τα δεκτυλικά τους αποτυπώματα. Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι έχουν μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλες χώρες Το 86% των ε, ε, ανθρώπων αυτών μεταβαίνει τελικά και σε άλλη χώρα Θα μπορούσε κανείς δηλαδή να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί μετεγκαθίστανται από την Ιταλία και την ε, ε, Ελλάδα σε μια άλλη χώρα, αλλά από εκεί και πέρα διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν και να συνεχίζουν τα ταξίδια τους και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, Βρετανία, Σουηδία. Για τα hot spot, είναι γεγονός ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι ε, καταστροφική, είναι ε, αποτρόπαιη και αυτό δεν είναι ε, fake news, δεν είναι ψευδείς ειδήσει. Το, το αποδεικνύουν οι εικόνες που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση και στις ειδήσει. σε ό,τι αφορά την κατανομή ανθρωπίνων πόρων, να το πω ήπια είναι κάθε άλλο παρά ιδανική. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι απαραίτητοι πόροι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα hotspot. Όσον αφορά τις επιστροφές, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αποδεικνύει ότι η επιστροφή στην πραγματικότητα είναι μια ιδεατή, μια επιθυμητή κατάσταση ε, χωρίς όμως να ε, εφαρμόζεται και να υλοποιείται στην πράξη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πρέπει να επιστραφούν δραπετεύουν, δραπετεύουν μέσω συγκεκριμένων οδών και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις όσον αφορά τους παράνομους ε, μετανάστες είναι φυγάδε. Παραθέτω τα λόγια της ίδιας της ειδική έκθεσης. Η απέλαση παράνομου μετανάστη κοστίζει 1890 ευρώ ε, σε κανονικό αεροπλάνο το 43% των θέσεων αυτών των αεροπλάνων που ναυλώνονται δεν καλύπτεται, ενώ στο 35% των ε, περιπτώσεων πρόκειται για συνοδευόμενα άτομα. Ενώ πολλοί ε, μετανάστες που έχουν απελαθεί, που έχουν επιστραφεί, τελικά επιστρέφουν στην Ένωση από άλλους δρόμους, από άλλες οδούς. Όλα αυτά αποδεικνύουν την καταστροφική κατάσταση και την επιτακτική ανάγκη να αναλυφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα εντάσσονται σε μια τελείως διαφορετική λογική. Και εδώ ε, περιλαμβάνει και σχετικές συστάσεις η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Εναπόκειται βεβαίως στην ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, να προστατεύουν τα σύνορά τους και κατά συνέπεια τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι αιτούντες άσυλο δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραμένουν να διαμένουν στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση και η επεξεργασία των αιτήσεών τους. Ξαναλέω, έως ότου ληφθεί μια οριστική απόφαση, οι άνθρωποι αυτοί έχουν με βάση το τρέχον καθεστώς το δικαίωμα να, ε, να μετακινούνται ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα άλλο, ένα διαφορετικό σύστημα επιστροφών, γιατί είναι πραγματικά απαράδεκτο να μπορεί κανείς να ε, μετακινείται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς κανέναν κανόνα. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είναι μέλη του χώρου Σέγγεν, κάτι που αποτελεί ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι αυτών των χωρών μπορούν να μεταφέρουν ε, να μετακινούνται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο αφού περάσουν έλεγχο διαβατηρίων το έχει ζήσει και η κυρία Κρέτσου. Δεν μπορεί να ισχύουν λιγότερο σοβαροί κανόνες, λιγότερο αυστηροί κανόνες για τους παράτυπους μετανάστες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Κρέτσου και μετά γονά. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι σκιώδης. Ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο και τον εισηγητή μας για την ε, πολλή δουλειά. Πολύ σημαντική ειδική έκθεση. Για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σωστά τόνισε ο εισηγητής. Τα τελευταία χρόνια η Ένωση έχει δει μια πρωτόγνωρη ένα πρωτόγνωρο κύμα μεταναστεύσεων τεράστιος αριθμός αιτήσεων ασύλου με κορύφωση το 2015 όπου ένα εκατομμύριο, πάνω από ένα εκατομμύριο επεδίωξαν να κάνουν αυτό το τόσο δύσκολο ταξίδι μέσω της θαλασσίας οδού. Το 2014-2020 έχουμε δαπανίσει 160 εκατομμύρια αλλά οι προκλήσεις και το γεγονός ότι μας εξέπληξε αυτό το κύμα μετανάστευσης έχουν ως αποτέλεσμα ότι αυξήθηκε η χρηματοδότηση και είναι 1,1 στο δισεκατομμύρια στο προπολογισμό 19. Λυπάμαι που το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι είναι μεγάλη η διαφορά μεταξύ στόχων και αποτελεσμάτων παρά το ότι αυξήθηκαν οι δυνατότητε στην Ιταλία και την Ελλάδα, διότι η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι δύο χώρε που λαμβάνουν τι περισσότερε χρηματοδοτήσει από το Ταμείο αυτό. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή των διαδικασιών στην Ιταλία και την Ελλάδα εξακολουθούν να καθυστερούν πολύ, όπως σας είπε μόλις ο εισηγητής. Ποιοι είναι οι λόγοι γι' αυτό. Είναι ότι υπάρχει ανεπαρκές δυναμικό στα κέντρα υποδοχής, δύσκολη η συνεργασία με τα κράτη προέλευσης και το γεγονός ότι μόλις ληφθεί η απόφαση επιστροφής τους, ορισμένοι μετανάστες εξαφανίζονται. Δύο ερωτήσεις. Αυτές οι αδυναμίες εφαρμογής των στόχων μας στην Ελλάδα και την Ιταλία οφείλονται σε ανεπαρκές ε, νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ή επειδή δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμες λύσεις που έχετε εντοπίσει για να αντιμετωπιστούν οι στενώσεις. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλές οι πέντε συστάσεις του συνεδρίου. Και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουν τις συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούνε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόιτς ανέφερε εντυπωσιακά στοιχεία ξέρουμε τη γνώμη που έχει ο Βίκτορ Όρμπαν έχει δημιουργήσει μια σειρά από συστήματα που σημαίνει ότι πρόκειται για άτομα και για κυκλώματα που έχουν να κάνουν με λαθρεμπόριο οπλών ναρκωτικών και με άτομα που έχουν να κάνουν δικτατούρα, με δικτατορία. Δεν ξέρω σε ποιου ε, υπερασπιστέ τη μετανάστευση που αναφέρεται ο κύριο Ντόιτς. Ο Όρμπαν και όλοι οι γύρω του κλέβουν τη χώρα μας και αποτελούν κίνδυνο για την ε, δημόσια ασφάλεια. Με τη συνεργασία του κύριου Όρμπαν μπαίνουν διάφοροι τύποι που έχουν τέτοιο παρελθόν και αυτό είναι ένα σοβαρό στοιχείο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κάτι άλλο σοβαρό. Ένα πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Γκρουεύσκη τη Μακεδονία. Ο Όρμπαν και η κυβέρνησή του, που ξέρουμε ότι είναι διακινητή ατόμων. Αυτό το άτομο το ε, δέχονται στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Όρμπαν. Και μετά εξακολουθούν να μιλάνε για... και να καταγγέλουν τους και να καταγγέλουν άλλους για φίλους της παράνομης μετανάστευσης. Η κυβέρνηση του Όρμπαν και το κόμμα του, ο ίδιος ο Όρμπαν είναι υπεύθυνοι για τέτοιες περιπτώσεις ε, χιλιάδες άτομα που έχουν ε, τέτοιο εγκληματικό παρελθόν και που τους έχουν δεχθεί στην Ουγγαρία και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. και μπορούν μετά να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την άδεια διαμονής που τους δίνει ο Όρμπαν. Έτσι η Ουγγαρία πρέπει να καταλάβει τι κάνει. Για το ελεκτικό συνέδριο θα ήθελα να πω το εξής. Σας συστήνω να δείτε πού είναι αυτές οι υπεράκτες εταιρείε που κάνουν αυτές τις ε, διαδικασίες. Υπήρξαν και αποφάσεις ουγγρικών δικαστηρίων που καταδίκασαν τον Όρμπαν και τον κύκλο του για αυτά που κάνουν μέσω υπόπτων συναλλαγών. Δεν έχουν ελεγχθεί όλα αυτά. Όλα αυτά τα άτομα που μπορούν ανα πάσα στιγμή να μπουν και να βγουν στο, στην Ένωση. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα ήθελα να κάνουμε τώρα ενδοουγγρικές συζητήσεις. Είναι ευρωπαϊκό θέμα αυτό. Οπότε αγαπητέ Στανφυρούνεν, αν ε, έχετε στοιχεία που να είναι ενδιαφέροντα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας παρακαλώ να τα στείλετε για να τα διερευνήσει. Γιατί εδώ στην Επιτροπή μας ε, δεν θέλουμε τώρα να κάνουμε συζητήσεις για εσωτερικά θέματα της Ουγγαρίας. Δεν νομίζω πως είναι κατάλληλος χώρος. Ο κύριος Πέξα. Ευχαριστώ πολύ. Να αντιδράσω κι εγώ σε αυτά που είπε ο κύριος Ντόιτς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές λέτε συνεχώς ότι είναι πρόβλημα η παράνομη μετανάστευση η παράνομη μετανάστευση κανένα άτομο δεν είναι παράνομο κανένα δικαστήριο δεν λέει ότι κάποιος είναι παράνομος Συγγνώμη, κανένα δεν είναι παράνομο εάν δεν έχει διαπιστώσει ένα δικαστήριο ότι είναι παράνομο. Άρα είναι θέμα κράτου δικαίου. Το κράτο δικαίου είναι η βάση του ευρωπαϊκού μα πολιτισμού και πρέπει να τηρούμε του κανόνε του. Η συζήτηση αυτή για τι επιστροφέ βεβαίω είναι σημαντική, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έρχονται σε μας Δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι και επαρκείς δυνατότητες αντιμετώπισης ε, των ατόμων αυτών χωρίς καθυστέρηση. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Και αυτή είναι η ερώτησή μου. Εάν λειτουργεί σωστά το σύστημα εξέτασης ετοιμάτων ασύλου. Εκεί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και εκεί θα πρέπει να βρούμε και λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Έπινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά τις, ε, τα χρυσά διαβατήρια. Θα ήθελα να ρωτήσω το Ελληνικό Συνέδριο αν έχει ερευνήσει το φαινόμενο αυτό. Όπως γνωρίζετε ενδεχομένω, η Μάλτα εισήγαγε το 2014 ένα σύστημα το οποίο επέτρεπε σε ανθρώπους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν την υπηκότητα της Μάλτας δηλαδή η ευρωπαϊκή υπηκότητα και πρόσβαση στη ζώνη Σέγγεν, πληρώνοντας 650.000 ευρώ σε εθνικό ταμείο ή αγοράζοντας περιουσία ή μετοχές. Το 2017 η, η Μάλτα εξέδωσε 1.400 διαβατήρια σε πλούσιους ανθρώπους κατά κύριο λόγο από τη Μέση Ανατολή και την Ασία και ένας από τους κινδύνους που περιλαμβάνει αυτή η οδός μετανάστευσης είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους από τα ανώτερα στρώματα ε, της κοινωνίας, κάτι που μπορεί να ε, δώσει τη δυνατότητα σε εγκληματίες ή ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και απευθύνω αυτό το ερώτημα στον κύριο Πρίνκατ. Γιατί μιλάμε για μια χώρα την οποία γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά. Πρόκειται για ένα σημείο εισόδου ε, εγκληματιών. Ε, εδώ ενώ ε, ταυτόχρονα στη Μάλτα διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση δολοφονίας της κυρίας Γκαλήθια. Οπότε το ελληνικό συνέδριο θα ήθελα να ρωτήσω ποια, ποια θέση έχει για αυτό το ζήτημα. Ε, η πρόεδρος ρωτά αν ο μιλητής αν, ανέφερε 400.000 διαβατήρια. Όχι, διορθώ, λέει ο, ο μιλητής, 1.400 διαβατήρια έχει εκδώσει η Μάλτα. Ναι, ωραία. Να δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Α, ο κύριος Κούς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ένα πολύ σύντομο ερώτημα θέλω να θέσω. Ε, διαπίστωσα ότι η, καταρχάς να, εκθέσω, να ευχαριστήσω το Ελληνικό Συνέδριο για την έκθεση, αλλά βλέπω ότι ασχολείται κυρίως με τα hot spots που δημιουργήθηκαν στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Γιατί δεν ε, εξετάσατε και ε, τα hot spots στην Θέουτα και τη Μελίγια, ε, αυτούς τους θύλακες, όπου επίσης υπάρχουν ε, hotspots. Και τι συμβαίνει με τη Μάλτα, γιατί ε, δεν ε, ε, εξετάστηκε και αυτή η χώρα στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ και με αυτό δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπρίνκατ για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και όλους εκείνους που έλαβαν το λόγο με ερωτήσεις. Καταρχάς επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι εγώ εκπροσωπώ το ελεγκτικό συνέδριο εδώ, με μια ιδιότητα την οποία ε, καλύπτω εδώ και τέσσερα χρόνια και είμαι εδώ για τις ειδικέ εκθέσεις για το άσυλο, την ε, επανεγκατάσταση και τις επιστροφές ε, που έχουν συγκεκριμένο πεδίο. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούν τις εκθέσεις και ελπίζω να δώσω τις ε, απαραίτητες πληροφορίες. Όσον αφορά την παρέμβαση του κ. Ντόιτς, είναι απόλυτα σαφές ότι οι αρχές ε, έφεσης ε, παραβλέπονται και συμφωνώ μαζί σας. Και εγώ είπα ότι εκ παραλήλου, όχι αντικαθιστώντας το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, θα πρέπει εκ παραλήλου να επισκέφτονται και αυτοί τα hot spot. Εγώ επισκέφτηκα και τη Σάμο και τη Μεσίνα και επιβεβαιώνω ότι η κατάσταση στα hot spot ε, είναι ε, φρικαλέα, οι, οι είναι αποτρόπες, ε, ακόμα χειρότερες από την πρώτη διερευνητική στολή που έγινε το 2018. Και το αποτέλεσμα για τις επιστροφές, συμφωνώ, είναι ανησυχητικό, ιδιαίτερα ανησυχητικό θα έλεγα, και στην έκθεση θα δείτε ότι στη σελίδα 58 δεν δώσαμε ένα μόνο λόγο, αλλά βρήκαμε 8 λόγους για τις ελλείψεις αυτές. Έχουν υπάρξει επικρίσεις για την αποτελεσματικότητα ή μάλλον την εγκυρότητα κάποιων πολιτικών, όχι την αποτελεσματικότητα. Και παρά το γεγονό ότι εκτιμώ ότι δεν ε, ε, επισερχόμαστε εμεί στα υπέρ και τα κατά ενό στόχου, αυτά ε, είναι αρμοδιότητα των ηθινόντων, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κοινοβουλίου που εποπτεύει. Ε, εμείς κοιτάμε να δούμε κατά πόσον ο στόχος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε εμείς ή όχι με το στόχο, έχει επιτευχθεί. Και αυτό που κοιτάζουμε να δούμε και ακόμα και ε, για αυτούς οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση για τους στόχους ε, και τα τελικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν. Νομίζω ότι η έκθεσή μας δείχνει σαφώς ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε αλλαγές για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και παρά το γεγονός ότι συμφωνώ ότι κάποιος από τους παριστάμενους ε, προσπάθησε να με υποχρεώσει να πω ποια θα ήταν τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία θα αποτελούσαν προτεραιότητα στους όρους που θέσαμε, πρέπει να σας πω ότι ειλικρινά, κατά την άποψή μας, και οι πέντε συστάσεις είναι εξίσου σημαντικές ε, και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για το ΕΑΣΟ τώρα, το Ίδρυμα Σύλλου, εκεί διαπιστώσαμε κάποιες ε, ελλείψεις ε, και αδυναμίες και να σας παραπέμψω στην σύσταση παριθμών 3, η οποία σαφέστατα λέει ποιες είναι οι αδυναμίες και επίσης ποιες είναι οι συγκεκριμένες συστάσεις ε, που σχετίζονται με αυτά και πιο συγκεκριμένα σύσταση παριθμών 5. Όταν παρουσιάσαμε την έκθεση και όταν ε, ε, μιλήσαμε με τα μέσα ενημέρωσης και επισκεφτήκαμε ε, κάποιες χώρες μέλη, γιατί έχουμε αφήσει έξω την Ισπανία και τη Μάλτα από την εξίσωση. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία και η Μάλτα δεν ήταν εντός του δικού μας του πεδίου. Ε, μπορεί να υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν τη Μάλτα, αλλά θα πρέπει να ρωτήσουμε τη Μάλτα όταν βλέπουμε το θέμα της μετανάστευσης. Ε, και τους είπα ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τη δική μου την υπηκότητα που είμαι Μαλτέζος. Εγώ είμαι εδώ πρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου. Επιλέξαμε την Ελλάδα και την Ιταλία, γιατί αυτή ήταν η εντολή που μας έδωσε σαφέστατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια μιας μελέτης που είχε γίνει από τον... Ε, ε, εκλειπώντα πλέον ε, Σουηδό εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου όταν έγινε η αρχική σύσταση και δείχνει ότι και το Κοινοβούλιο ένιωσε ότι υπάρχει μια αίσθηση κατεπήγοντος ε, και γι' αυτό ζήτησαν μία επιπλέον έκθεση αμέσως και δεν περιμέναν τρία-τέσσερα χρόνια για να υπάρξει επόμενη έκθεση. Το ίδιο το Κοινοβούλιο δηλαδή διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να επέμει το πρόβλημα και έπρεπε κάπως να κάνουμε μία επιπλέον έκθεση για να τα δούμε. Προέκυψε δε σαφέστατα ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι χώρες μέλη που πλήττονται περισσότερο από την ε, μετανάστευση από το 2015 και όσον αφορά τις αφήξεις και όσον αφορά τις αιτήσει ασύλου. Όπω σα είπα και προηγουμένω, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι μόνε χώρε που ζήτησαν και έχουν εφαρμόσει συγγνώμη, μέχρι τώρα την προσέγγιση των hot spot και το 2015 γνωσήθηκε και μια πολύ καλή έκθεση και έγινε και αποδεκτή από το Κοινοβούλιο αλλά το Κοινοβούλιο ήθελε να παρακολουθήσει τις συστάσεις του ελέγχου μας αυτού. Επομένως, εμείς, αντί να διεξάγουμε μια νέα ε, διαδικασία ελέγχου, εξετάσαμε κατά πόσον ήταν αποτελεσματικές ή όχι οι συστάσεις που κάναμε το 2017. Η Ελλάδα και η Ιταλία ε, είναι και αυτά μεταξύ των κρατών μελών, με την, ε, εκτός από την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, που λαμβάνουν και επιχειρησιακή στήριξη από την ΕΑΣΟ. Και επίσης υπάρχουν και δύο ακόμα σημαντικές πτυχές. Ε, τα προγράμματα επίκουσας μετεγκατάστασης που έγιναν στην Ελλάδα και στην Ιταλία και το γεγονός ότι η Ιταλία και η Ελλάδα είναι αυτές που υποδέχονται ε, και λαμβάνουν μάλλον ε, την κατεπίγουσα χρηματοδότηση. Αυτά είχαν να απαντήσω αν δεν κάνω λάθος. Να επανέλθω όμως στο αρχικό ερώτημα για το κατά πόσον είναι λογικό να χρειάζεται τόσος χρόνος για να εξετάσει κάποιος ε, μία αίτηση ασύλου. Για την Ελλάδα να σας παραπέμψω στο σχήμα 17 και τις παραγράφους 112 με 114. Είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτας εργασίας για τις ε, ε, αρχές τις οποίες ασκείται έφεση μετά την απόφαση ε, ε, ασύλου, γιατί δεν η Ιταλία υπάρχει αντίστοιχη ε, διαπίστωση. Χρειάζεται πολλής χρόνος για τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων ε, ε, ασύλου και στο στην επόμενη παράγραφο λέγεται σαφέστατα ότι η τελεσίδικη απόφαση μπορεί να διαρκέσει και τέσσερα χρόνια. Συμφωνώ απολύτω ότι πολλέ χώρε μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι απολύτω απαράδεκτο και απάνθρωπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς επιδεικνύουμε μεγάλο σεβασμό σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου, ανεξάρτητα από την υπηκότητά τους και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι το έργο που επιτελούν είναι εξαίρετο και ότι εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που θα ήθελε κάποιος να θέσει. Ίσως ε, η Κομισιόν θα ήθελε να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ. Ναι. Όχι για να υποβάλω ερωτήματα, αλλά για να σας υποβάλω κάποια σχόλια. Με χαρά βεβαίως. Ξεκινώ κι εγώ με την ίδια παρατήρηση που έκανα και για την προηγούμενη έκθεση. Ότι θέλω να ευχαριστήσω δηλαδή το υπεύθυνο μέλος του Ελληνικού Συνέδριου, τον κύριο Μπρίνκατ και το επιτελείο του που συνεργάστηκε μαζί μας για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης και σε αυτή την περίπτωση είχαμε εξαιρετική συνεργασία και πρέπει να σας πω ότι έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλές ανταλλαγές πληροφοριών γιατί πράγματι, όπως είπατε κι εσείς, η έκθεση καλύπτει ένα σχετικά στενό φαινομενικά ε, πεδίο στην πραγματικότητα όμως ε, επικεντρώνεται στο, στον πυρήνα της ε, εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής και πολλές πτυχές που συνδέονται με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής στο μέλλον. Στο μέλλον. Υπάρχει λοιπόν μια εξαιρετική πραγματολογική περιγραφή της κατάστασης έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά τις συστάσεις, αν συνυπολογίσει κανείς και τις υποσυστάσεις, ε, ο αριθμός τους είναι και πολύ μεγάλο και είναι πολύ χρήσιμε οι συστάσεις, ακριβώς γιατί αποτελούν και μια συνέχεια προς την πρώτη έκθεση που είχε συνταχθεί με αντικείμενο τα hotspot. Σας ευχαριστώ λοιπόν και αναγνωρίζω όπως και στην προηγούμενη έκθεση το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ θετικές ε, παρατηρήσεις, ιδίως ε, διότι αναγνωρίζεται ένα συνεχές. Διαπιστώνεται ανάμεσα στις δύο εκθέσεις ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, ιδίω όσον αφορά την ικανότητα των Ιταλικών και Ελληνικών αρχών, τις δυνατότητες που έχουν οι αρχές αυτές για την διεκπαιρέωση αιτήσεων, όσον αφορά τη συνεργασία ε, όσον αφορά τι συστάσει μάλλον του 2017, οι περισσότερε από αυτέ έχουν εφαρμοστεί ή βρίσκονται στο στάδιο τη εφαρμογή. Ότι η καταχώρηση δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, μεταναστών στα hotspot έχει βελτιωθεί πολύ και μεγάλος αριθμός, μεγάλο μερίδιο, μεγάλο μέρος των ε, ετούντων άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί. Επομένως, οι εξεταστήσει δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιταλία και στην Ελλάδα ε, προσδιορίστηκαν με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και έτσι περάσαμε στην ε, νέα ε, φάση των συστάσεων, οι οποίες έχουν γίνει πλήρως αποδεκτές από εμάς και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τις εφαρμόσουμε. Στο πλαίσιο βεβαίως και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας θα υποστηρίξουμε και θα διευκολύνουμε την εφαρμογή αυτών των συστάσεων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και, και σε συνεργασία με τους οργανισμούς. Έχουν άλλωστε γίνει και σχετικές συζητήσει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι παράγοντες της διαδικασίας θα εφαρμόσουν και θα υλοποιήσουν αυτές τις συστάσεις με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. Έγινε ένα σχόλιο σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες άξεις, πράξεις, δράσεις. Ε, θυμήθηκα λοιπόν ότι προς το τέλος της ε, θητείας της προηγούμενης Κομισιόν υπήρχε ένα θυματολόγιο για τη μετανάστευση που πρότεινε η Κομισιόν στην αρχή περίπου της μεταναστευτικής κρίσης όπου προτείνονταν συγκεκριμένα συγκεκριμένα βήματα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να ε, υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης. Αυτό τότε είχε γίνει με την, ε, με την πεποίθηση ότι η μετανάστευση είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο και ε, έγινε με ε, καλή πρόθεση προκειμένου για το, ε, για πώς θα πρέπει να, διαχειριστούμε την μετανάστευση τα επόμενα χρόνια. Ε, είδατε όμως ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι έγιναν ξαφνικά άμεση στόχοι, όπως είναι η δημιουργία επιχειρησιακών ικανοτήτων, όπως ήταν η δημιουργία των hotspot, γιατί αυτό ήταν, αποτέλεσε από τη μία μέρα στην άλλη άμεσο στόχο, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο, προκειμένου να βοηθωθούν τα κράτη-μέλη που ήταν στην πρώτη γραμμή της υποδοχής των μεταναστών και που αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα για τη διαχείριση της ε, μεταναστευτικής κρίσης. Για πρώτη φορά λοιπόν καταφέραμε και ε, εξασφαλίσουμε συνεργασία οργανισμών και κρατών μελών. Αυτές οι, αυτές, αυτές οι βραχυπρόθεσμες δράσεις ε, λοιπόν, έγιναν άμεσες δράσεις ξαφνικά. Το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο μάλλον συνέβη με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις. Πράγματα τα οποία σχεδιάζαμε να τα κάνουμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, τελικά αναγκαστήκαμε να τα επιταχύνουμε, να τα κάνουμε πολύ πιο γρήγορα και αυτό ε, επίσης νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Όπως είπα λοιπόν, εμείς θα ε, παρακολουθήσουμε τις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που απευθύνονται στην Κομισιόν. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ιταλία ως προς την εφαρμογή αυτών των συστάσεων και θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια η αποφασιστική δράση της Κομισιόν αλλά και η συλλογική δράση που ανελήφθη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βελτίωσε σημαντικότατα την ποιότητα της διαχείρισης της μετανάστευσης. Σήμερα πια είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν ε, ώστε να παράσχουμε πρακτική και οικονομική χρηματοδοτική βοήθεια προς την ε, Ελλάδα και την Ιταλία και σε όλες τις χώρες που δέχονται μεγάλες πιέσεις από μεταναστευτικές κινήσεις. Αυτή η προσέγγιση των hot spot η οποία, η οποία θεσπίστηκε, αν θέλετε, δημιουργήθηκε στην αρχή της μεταναστευτικής κρίσης, βοήθησε στη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζαμε εκείνη την περίοδο. Μεγάλο τμήμα της έκθεσης επικεντρώνεται στην εφαρμογή της ε, πολιτικής μετεγκανάστασης, τον πολιτικό σχεδιασμό αυτής και, τον, ε, και την εφαρμογή της. Και η μετεγκατάσταση ήταν πραγματικά μια απόδειξη της ευρωπαϊκής Ελληνική, Γιατί αν λάβει κανεί υπόψη του τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην, ε, στις αποφάσεις στις οποίες βασίζεται η μεταγκατάσταση ε, έχουν ε, μεταγκατασταθεί πάνω από 100.000 άνθρωποι στη βάση των πολιτικών και των κριτηρίων που είχαν καθοριστεί με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται και μια δίκαιη κατανομή των βαρών στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρότι είναι εθνική αρμοδιότητα η πολιτική για τις επιστροφές και η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η υποστήριξη της Κομισιόν και των οργανισμών ε, αποτέλεσαν κρίσιμης σημασίας, ε, ζωτικής σημασίας ε, στοιχεία για την βελτίωση της κατάστασης και για την υποστήριξη που παρέχεται προς, την, ε, προς τα κράτη-μέλη που δέχονται πιέσεις. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή την επιχειρησιακή και χρηματοδοτική στήριξη σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη ώστε να ενισχύεται και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Για, τα, για τους μηχανισμούς Θέλω να πω το εξή. Όταν μιλώ για κριτήρια και μιλώ για το 100% των, των κριτηρίων, αυτό σημαίνει ότι 35.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και την Ιταλία που ε, έχριζαν διεθνούς προστασίας έχουν μεταγκατασταθεί. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, αποδεικνύει την σημασία και την αποτελεσματικότητα των κριτήριων που ε, θέσαμε. Για τι διαδικασίε ασύλου και μετανάστευση είναι προφανέ ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις τελικές και ελληνικέ αρχές. Και να πω ότι η τρέχουσα κατάσταση, η οποία βελτιώνεται πρέπει να πω, ε, θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο των εργασιών μας και της συνεργασίας μας με τις Ιταλικές και Ελληνικές Αρχές και θα επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Στην ε, Ελλάδα μάλιστα έχει ψηφιστεί και νέα νομοθεσία η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από, τις, ε, από 1η Ιανουαρίου και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα για την βελτίωση της κατάστασης. Όσον αφορά τις επιστροφές, μια αποτελεσματική ε, και ανθρωπιστική πολιτική επιστροφών ε, βασίζεται στην αρχή ότι εκείνοι που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα την λαμβάνουν, εκείνοι που διαπιστώνεται ότι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας θα επιστρέφονται. Η κατάσταση βεβαίως δεν είναι ιδανική, το ξέρουμε. Το ποσοστό των επιστροφών εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Θα συνεχίσουμε όμως το έργο που ξεκινήσαμε με το σχέδιο δράσης, με τις συγκεκριμένες συστάσεις του 2019 και με τις προτινόμενες ε, αναθεωρήσεις, τις συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου και την ε, συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης. Νομίζω ότι συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο αυτές εκθέσεις καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα ε, πτυχών της, ε, της μετανάστευσης ε, πρόκειται για φαινόμενα τα οποία αξιολογήθηκαν και εκτιμήθηκαν από το Ελληνικό Συνέδριο, για διδάγματα που αντλήθηκαν και που μετουσιώθηκαν σε συστάσεις, τις οποίες και θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε και αυτό αποδεικνύει με τη σειρά του ότι υπάρχει μια τεράστια και πολυσχηδής εικόνα ε, η οποία απαρτίζεται από πολλές επιμέρους εικόνες και που μας ε, ε, αποδεικνύει ότι χρειάζεται συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, από το, από το ευρωπαϊκό έως το εθνικό επίπεδο και βεβαίως συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά από πλευράς Κομισιάν. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστούμε το ηλεκτρικό συνέδριο για την εργασία του, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τυπικές αυτές οι ευχαριστίες. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι πιστεύω Καλό είναι να ρωτάμε το Συμβούλιο, καλό είναι να ρωτάμε διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και τις ε, συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, αλλά πρέπει να διαπιστώσουμε ένα λάθος. Το Ελεκτικό Συνέδριο κάνει μια σοβαρή και τεκμηριωμένη εργασία. Είναι σαφές αυτό. Και μας λένε τα πράγματα όπως είναι. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό και μας έδειξε η έκθεση αυτή μια κατάσταση πολύ ανησυχητική. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας της συζήτηση. Δεν το λέω αυτό γιατί θέλω να περασπιστώ το συνέδριο που δεν χρειάζεται να το περασπιστώ εγώ. Μπορούμε να συζητήσουμε και να εξαγάγουμε και διαφορετικά απορίσματα, αλλά δύο στοιχεία πρέπει να είναι αδιαφυσβήτητα. Εν σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και το σημείο αφετηρίας λέγω λοιπόν ότι είναι ότι υπάρχει μία και υπήρξε μία μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη και γίνεται μια συζήτηση πολύ σοβαρή τώρα για το πώς να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι τώρα η στιγμή να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση. Αυτό πρέπει να πούμε σαφώς είναι ότι ανεξάρτητα από το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, η αντιμετώπιση αυτή πρέπει να είναι αποτελεσματική. Και η εργασία του Λογικού Συναδρίου καταδεικνύει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής επαρκώς αποτελεσματική. Ορισμένοι λένε βέβαια ότι ναι μεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που περιγράφει το ελεκτικό συνέδριο Ορισμένοι μπορούν να λένε λοιπόν ότι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πρέπει να αλλάξουμε τους στόχους ή να αλλάξουμε τις μεθόδους. Αυτές τις δυνατότητες έχουμε. Έτσι πρέπει να συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με βάση αυτή την τόσο χρήσιμη βάση. Και σε ευχαριστώ όλου. Ευχαριστώ πολύ και πρόεδρο, τον εισηγητή μα και ευχαριστούμε όλου ιδιαίτερος τον κύριο Μπρίκατ, μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου και την Επιτροπή για την εξαντλητική παρουσία μας έκανε. Το θέμα αυτό θα μας ε, απασχολήσει και στο μέλλον γιατί έχει και επιπτώσεις ε, στους πόρους της Ένωσης, στους πόρους των φορολογουμένων. Έτσι νομίζω ότι σολομοντίως μπορεί να ολοκληρώσω του, τη συζήτηση. Ξέρετε ότι πάντα ε, η ιστορία καταδεικνύει ότι τιμωρούμε πολύ συχνά τον αγγελιοφόρο και όχι αυτόν που μας φέρνει τις κακές ειδήσει και όχι αυτόν που έχει προκαλέσει την κακή κατάσταση. Ευχαριστώ λοιπόν για τη σκληρή εργασία σας και την ε, ετοιμότητά σας να δεχθείτε και αδικαιολόγητη κριτική. Λοιπόν, καλή επιστροφή στο Λουξεμβούργο, με τρένο υποθέτω. Στις 16-12 του θα έχουμε μια ειδική συνεδρίαση στο Στρασβούργο και κλεισμένων των θυρών όπως το συζητήσαμε με τον κύριο Επίτροπο. Για να συνεχίσουμε τη ζήτηση και κλεισμένων λοιπόν και σε ευχαριστώ πολύ. Λήξη της συνεδρίας. Yes, yes, yes.